Ε, Παρακαλώ να καθίσετε. Θα συνεχίσουμε τη συνάντηση. Να σα ενημερώσω ότι για την Επιτροπή μετέσχων στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Συνεργασία στην Ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Σεγκόβια στην Ισπανία. Μετά τη, με βάση την καλή παράδοση που έχουμε εδώ και κάποια χρόνια, η Ισπανική Προεδρία είχε καλέσει αυτή την άτυπη συνάντηση την πρόεδρο της Επιτροπής μας για το Κοινοβούλιο και τον συνάδελφο κ. Λίμισε ως συμπρόεδρο της, της Ισομερούς ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ ΕΕ. Στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν ε, τα εξή θέματα. Η παρουσίαση του προγράμματο εργασία από τον Επίτροπο Πίμπαλ. η προετοιμασία τη Συνόδου Κορυφή τη Νέα Υόρκη του ΟΗΕ για του στόχου τη χιλιετία, η αποτελεσματικότητα τη βοήθεια, ο καταμερισμό εργασία, ο κατακαιρματισμό τη ενίσχυση και ο πολλαπλασιασμό των δωρητών, η καλή διακυβέρνηση στον τομέα, στο φορολογικό τομέα για την ανάπτυξη, ένα σημείο για το οποίο ε, είχε προσκληθεί και υφυπουργός ανάπτυξης της Νορβηγίας και για το οποίο είχε κληθεί να κάνει και μία παρουσίαση. Ο διατλαντικός διάλογος στον τομέα της συνεργασίας είναι ένα θέμα που εξετάσαμε με τον υπεύθυνο του USA των ΗΠΑ, κύριο Ρατζίβ Σαχ. Εξετάσαμε επίσης την κατάσταση στην ΑΕΤ ένα θέμα που συζητήθηκε παρό, της Επιτρόπου Γεωργίευα του κ. Ρατζίφ Σάχ για τις ΗΠΑ και του Εντμό Μιουλέ, ε, αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ειδικού απεσταλμένου για την IT. Ήταν μια μεγάλη μερίσια διάταξη. Δουλέψαμε από τι 9 το πρωί μέχρι τι 11 το βράδυ. Δεν ε, μπορώ να σας πω πλήρως το τι συζητήθηκε. Απλά να σας πω ότι απογοητεύτηκα κάπως από τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής ιδίως δε από την απουσία μέσων που θέτουν τα κράτη-μέλη στη διάθεση της επίτευξης των στόχων της χιλιετίας. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Έξι από τα 27 κράτη δεν τηρούν τις υποσχέσεις που είχαν δώσει προς την διεθνή κοινότητα, μεταξύ αυτών η Γαλλία. Très triste de voir que on abandonne Επίσης, με λύπη διαπίστωσα ότι εγκαταλείπεται η ιδέα της επίτευξης των στόχων της ήλετίας και γίνεται επικέντρωση σε κάποιους στόχους και όχι στο σύνολο. Αυτό το βρήκα κάπως απογοητευτικό. Πιστεύω ότι οι υπουργοί συμπεριφέρονταν περισσότερο ως υπουργοί οικονομίας και όχι ως υπουργοί ανάπτυξης. Δεν, είχ, δεν έδειχναν τον απαιτούμενο φυσιασμό. Αυτή ήταν δική μου άποψη. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη προφανώ για τη διαχείριση του προπολογισμού. Βρίσκω όμω πραγματικά ενοχλητικό να αναλύουμε γιατί δεν επιτυγχάνουμε του στόχου τη ηλικία, ενώ δεν τηρούνται οι δεσμεύσει. Ε, για το 0,51. Πολλές χώρες έχουν ε, μόνο 0,20% του ΑΕΠ τους ε, στην ανακτησιακή βοήθεια. Τέλος πάντων, αν θέλετε, να σας πω σε ατομικό επίπεδο με περισσότερες λεπτομέρειες τις συζητήσεις. Έχει να κάνει κάποιες αναγγελίες η Επιτροπή, κάποιες ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε. Οι ερωτήσεις. Λάβαμε Μία ερώτηση προ την Επιτροπή για τη συνάντηση αυτή, η οποία βρίσκεται στο ενίο φάκελο, στον ενίο φάκελο των βουλευτών. Υπενθυμίζω ότι μόνο η συντάκτη τη ερώτηση εγώ δηλαδή, έχει το δικαίωμα να θέσει συμπληρωματική ερώτηση. Η ερώτηση βρίσκεται στο φάκελό σα. Δεν την διαβάσω λοιπόν. Η Επιτροπή έχει το λόγο για την απάντηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που θέσατε προς την Επιτροπή, όντως ε, παρακολουθούμε το προεκλογικό πλαίσιο στη Ρουάντα εκ του σύνεγγης. Επίσης έχουμε πληροφορηθεί για κάποια περιστατικά που έλαβαν χώρα πρόσφατα και που αφορούσαν ορισμένα μέλη τη αντιπολίτευση. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση και τη γενικότερα την προεκλογική περίοδο, η αντιπροσωπεία τη Ένωση και τα κρατη και με τα κράτη-μέλη προέβη σε μια σειρά διαβημάτων προ τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ρουάντα. Ε, το τελευταίο διάβημα ε, έγινε στι 11 Δευτέρου. Στην συνάντηση εκείνη συζητήθηκε το θέμα της καταχώρησης των πολιτικών κομμάτων εν ώψη των προεδρικών εκλογών και τον, για τα επεισόδια ε, της, που, ε, τις οποίες ήταν θύμα η υποψήφια κυρία Βικτουάρ Εγκαμπιρέ. Κατά τη διάρκεια του διαβήματος αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την χρήση των μεθόδων εκφοβισμού και της βίας κατά οποιοδήποτε υποψήφιου ε, στις εκλογές και επέμενε ιδιαίτερα στο δικαίωμα των υποψηφίων να καταχωρήσουν την υποψηφιότητά τους, να υπάρξει καταχώρηση πολιτικών κομμάτων, ελευθερία το λειτουργίας των πολιτικών ε, κομμάτων και γενικά ελευθερία προεκλογικού χαρακτήρα. Να σας πω επίσης ότι η Επιτροπή θα συναντήσει και συναντά στη Ρουάντα όλους τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να υποβάλουν ενδεχόμενα υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές προσπαθούμε να περάσουμε ένα γενικό μήνυμα ότι όλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Ιδιαίτερα τον, τον νομοθετικό πλαίσιο και τον εκλογικό κανονισμό. Επίσης προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε φράση που μπορεί να έχει προκλητικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάτε ότι η Ρουάντα είναι μια κόρα που ζει ακόμα σε μια ε, το ότι ε, κοινωνική και δεν θα έλεγα αθηνοτική κατάσταση, είναι σημαντικό να προχωρήσει σε ειρηνικές εκλογές και να προωθηθεί η λειτουργία πολιτικών κομμάτων που θα έχουν όραμα για το μέλλον και που θα προσπαθούν να μην χρησιμοποιήσουν τις εκλογές για να φτάσουν σε ένα διακανονισμό μεταξύ τους που μπορεί να δημιουργούσε κινδύνους για τη χώρα και να ξανά τα νοπά τραύματα της κοινωνίας της Ρουάντα. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εκλογική διαδικασία και στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου με την ε, Ρουάντα θα συνεχίσουμε, αν προκύψει, να θέτουμε το ζήτημα της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών ανοιχτών για όλους. Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι στις τελευταίες ε, βουλευτικές εκλογές είχε μεταβεί εκεί μια αποστολή, εκλογική αποστολή της Επιτροπής και κάποιοι βουλευτές μάλιστα με επικεφαλής τον κύριο Κάσμαν. Η Επιτροπή αυτή είχε προβεί σε μια σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της, ε, της εκλογικής διαδικασίας. Πολλές από τις συστάσεις αυτές ε, λήφθηκαν υπόψη και εφαρμόζονται, εισάγονται, ενσωματώνονται στον υποσυζήτηση νέο εκλογικό κώδικα που συζητείται τώρα τελευταία, αυτό το τελευταίο καιρό. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει βελτίωση και έχουμε αρκετή βεβαιότητα ότι η, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κάτω από γαλήνιους όρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Με, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγις τις εκλογές αυτές. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και ότι όλα τα προβλήματα και όλες οι παρενοχλήσεις που υφίστανται υποψήφοι της αντιπολίτευσης θα καταγράφονται από την Επιτροπή, η οποία θα επαγρυπνεί. Έβδομο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και η έννοια της επίσημης βοήθειας για ανάπτυξη συν. Η συνάδελφος κυρία Κέλλερ θα παρουσιάσει τις βασικές ε, ιδέες που περιλαμβάνει το σχέδιο έκθεσης της. Θα συζητήσουμε με βασικούς ε, συνομιλητές ε, από την Επιτροπή και από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης e-Concord θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο που σας έχει δοθεί για να μπορέσουμε να έχουμε και μια συζήτηση. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Μάντσερ που δεν έφτασε ακόμα, αλλά θα ξεκινήσουμε ακούγοντας πρώτα την κυρία Φραντσέσκα Κέλλερ. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνέβαλαν και τους ε, σκιώδεις ηγητές, στην ε, γραμματεία και όλους όσους με βοήθησαν σε αυτή την μακρά διαδικασία που ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική. Όπως ξέρουμε υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και συνέπειες, περιπτώσεις στην, στην ευρωπαϊκή πολιτική, στην αλληλεία, στις, στα πνευματικά δικαιώματα, στη μετανάστευση, στα οικονομικά, στα όπλα, στα υλικά, στις πρώτες ύλες κτλ. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και με την έκθεση προσπαθούμε όχι μόνο να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση πέριξ αυτών των προβλημάτων, αλλά και να επαναβεβαιώσουμε την δέσμευση του Κοινοβουλίου για την ε, εκπόνηση σωστών πολιτικών και να θέσουμε σωστά ερωτήματα για το πώ μπορεί τελικά να εφαρμοστεί αυτή η δέσμευση και πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την συνοχή των πολιτικών. Είναι σαφέ ότι αυτέ οι ασυνέπειε δεν μπορούν απλώ να εξαφανιστούν όταν αντιμετωπίζουμε ένα ή δύο, μια ή δύο περιπτώσει που είναι ίσω οι πιο ε, έκδηλε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα και όλες οι υπηρεσίες αυτών των θεσμικών οργάνων συνεργάζονται έτσι ώστε αυτές οι ασυνέπειες να μπορούν να, προληφθούν το... Ε, ε, στο μέλλον ε, στο πλαίσιο του άρθρου 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Λοιπόν, μερικές από τις προτάσεις μας. Η έκθεση ζητά σαφή... σαφείς δείκτες και συγκεκριμένα κριτήρια και προτείνει ότι οι ε, δείκτε για την ανθρώπινη ανάπτυξη θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Επίση, ε, υπάρχει μια, ε, ζητείται ένα μηχανισμό παραπώνων για, την, για τι πολιτικέ, για την συνέπεια και για την ανάπτυξη οι οποίες δεν ε, τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν ε, τεθεί. Επίσης, το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα μπορούσε να είναι το σωστό βήμα για να ε, υποβληθούν αυτά τα παράπονα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον εκπρόσωπο σήμερα, γιατί αυτός είναι, υποβάλλει την ετήσια έκθεση και έχει ερευνητικές αρμοδιότητες για την υποβολή ε, ίδια έκθεση πρωτοβουλία για προβλήματα που προέρχονται από του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη εντολή που έχει. Επίση, η έκθεση προ την Κομισιόν ζητά να δώσει ε, σαφή ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή Τη βοήθεια σε όλες τις αναπτυγισόμενες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην παρούσα συζήτηση για το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου που θα καθορίσει το πόσο ε, συνεπεί και συνεκτικές θα είναι στο μέλλον οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Ω καθήκον του Κοινοβουλίου προτείνω στην ετήσια έκθεση να ε, για την, ε, να προετοιμάζεται μια έκθεση για την αναπτυξιακή πολιτική από το Κοινοβούλιο. Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα που έχω υποβάλει στην έκθεσή ε, μου, αλλά είναι σημαντικό για μένα να ολοκληρώσουμε αυτή τη ε, διαδικασία, μόλις στην Ολομέλεια εγκριθεί αυτή η έκθεση, αλλά να συνεχίσουμε και να εργαζόμαστε ως προς αυτήν, γιατί η Επιτροπή μας μπορεί πραγματικά να είναι ένας ε, πολύ αυστηρός ελεγκτής και εντός του οίκου μας, αλλά και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό προετοίμασα μία λίστα ε, συστάσεων για το τι μπορούμε εμεί στα πλαίσια τη Επιτροπή μα να κάνουμε για να ενισχύσουμε την, ε, την, τη συνοχή των πολιτικών. Για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο εισηγητή για την ε, συνέπεια των πολιτικών. Αυτά όλα θα τα βρείτε στην έκθεση. Και έχουμε προτείνει επίσης να εγκρίνουμε μια διαδικασία όπου εσείς θα στέλνετε τις δικές σας προσθήκες, ε, τα κριτικά σας σχόλια, ε, ε, τα παραπονά σας, τις προτάσεις σας και θα τα παρουσιάζουμε στην επόμενη συνεδρίαση, έτσι από κοινού, για να βλέπουμε τι προτάσει υπάρχουν και να υπάρχει υποστήριξη αυτών στην Επιτροπή πριν προωθηθούν περαιτέρω. Αυτή είναι μια διαδικασία που βοηθά όλους μας να συμμετέχουμε και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις ώστε μετά από έξι μήνες ή ένα χρόνο να μπορούμε να επανέλθουμε και να δούμε πού τα πήγαμε καλά και πού όχι. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Διευθυντή τη Γενική Διεθνή Ανάπτυξη, ε, κ. Μανσερβή, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Κομισιόν, Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια. Γιατί αυτή η έκθεση είναι και αυτό το θέμα είναι από τα πιο σημαντικά το μέλλον των, ε, των ε, αναπτυξιακών πολιτικών. Συμφωνούμε λοιπόν ε, όχι μόνο στη σημασία αλλά και σε πολλές από τις, και με πολλές από τις συστάσεις που υπάρχουν στην έκθεση. Γιατί λέω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Καταρχήν γιατί θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Επομένως αυτό απαιτεί ενισχυμένη πολιτική δράση και έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το νέο μέτωπο της ε, αναπτυξιακής πολιτικής και αν θέλουμε αυτή η πολιτική να μην ε, καθορίζεται απλώς από την ε, αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να γίνει κάτι που θα είναι ο προπομπός όλων αυτών των διαδικασιών για την εκπόνηση πολιτικών. Η συνεκτική πολιτική είναι, πρέπει να είναι στον πυρήνα. Το καλωσορίζουμε λοιπόν, παρόλο που ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Δεύτερον, γιατί αυτή είναι μια καινούργια ατζέντα που έχουμε. Είναι ένα ε, υποπροϊόν, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι ένας τρόπος για να ενισχύσουμε την ε, ευρωπαϊκή δράση στον τομέα της ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να έχουμε απλώς μια πολιτική που θα, που θα ε, εφαρμόζεται σε επίπεδο κρατών μελών. Καλύπτει όλη την Ένωση. Επομένως, ταιριάζει πάρα πολύ καλά με, την, με τις υπόλοιπες πολιτικές και το τονίζω, τονίζω την, τη, σημασία της, ε, συνεκτικό, της πολιτικής γιατί μπορούμε έτσι να εξεύρουμε τομείς που θα μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο για να υπάρξει όντως αυτή η συνοχή. Το καλωσορίζουμε λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί και μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συγκεκριμένο, έχουμε, ε, έχουμε βρει πέντε βασικές προκλήσεις. Όχι τυχαία. Κλιματικές αλλαγές, ασφάλεια, μετανάστευση, εμπόριο και οικονομία και ασφάλεια των τροφίμων. Είναι ήδη οι τομείς που δείχνουν ότι χρειάζεται συνοχή. Δεν είναι απλώς πολιτικές μεμονωμένες, αποξενωμένες η μία από την άλλη. Είναι τομείς που μπορούν να τους δούμε σε πολιτικό επίπεδο μόνο αν τους δούμε στο σύνολο, το, στο σύνολο τους και με το σύνολο των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί ότι οι 12 τομείς και οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από το 2005 θα αντικατασταθούν, αλλά μπορούμε ε, να το κάνουμε με έναν τρόπο που ήδη θα δείξει ένα διαφορετικό, μια διαφορετική προσέγγιση. Όταν μιλούμε ας πούμε, για τα τρόφιμα, δεν μιλούμε μόνο για τη γεωργία, μιλούμε για πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να, μπορούμε να επενδύσουμε στην γεωργία, αλλά από την εμπειρία μας και τώρα με την διάμεση αναθεώρηση, δεν λέει ότι απλώ ενισχύουμε την ασφάλεια των τροφίμων, επομένω ενισχύουμε μόνο την ε, γεωργία, γιατί μιλούμε και για βασικέ ε, υποδομέ των αγορών. Μιλούμε ότι, ε, για το ότι πρέπει να, επι, να επενδύσουμε στην πολιτική και στα πρότυπα. Να επενδύσουμε, ας πούμε, στις περιφερειακές πολιτικές για τη διεύρυνση των αγορών. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να το πούμε. Βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε τους 12 στόχους που σας είπα που έχουμε θέσει. Και επίση, στον πυρήνα των όσων κάνουμε είναι το πρόγραμμα εργασία για, την πολιτική, για τη συνθηκή πολιτική για την ανάπτυξη. Έχουμε συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένου δείκτε για να μπορέσουμε να τη μετρήσουμε. Γιατί όντω είναι δύσκολο να, το, να χαράξουμε μια τέτοια πολιτική, αλλά είναι, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να, να εφαρμόσουμε μια δύσκολη πολιτική. Γιατί η πολιτική δράση και ο έλεγχο του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι πιο ενισχυμένο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε έναν ε, πίνακα κατάταξη για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και μετά να δούμε μεταξύ μα ε, τι έγινε και τι δεν έγινε και γιατί. Αυτό το πρόγραμμα εργασία θα μεταδίδεται, θα αποδίδεται, αποστέλλεται και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Επομένω, εμεί περιμένουμε ότι το Κοινοβούλιο θα αναλάβει ηγετικό ρόλο, γιατί αυτό απαιτεί ένα αλφα επίπεδο σχέσεων ε, ή διασύνδεσης με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί πολλές πρωτοβουλίες ξεκινούν από τα κρατημέλη Επομένως, ε, αυτό μπορούμε να το ε, διαχειριστούμε από κοινού με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης, για τους συγκεκριμένου μηχανισμούς που αναφέρονται στην έκθεση, για τον μηχανισμό αυτόν συγκεκριμένα της υποβολής παραπώνων, πρέπει να πω ότι δεν είμαι σίγουρος πως θα είναι χρήσιμος ένας τέτοιος μηχανισμός και πρακτικός, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι. Για παράδειγμα, το άρθρο 12 της Συμφωνίας Κοτονού αυτή είναι η θεσμική επίσημη ας απάντηση που μπορώ να σας δώσω, ότι δεν συμφωνώ πολύ, αλλά προσωπικά, αν με ρωτάτε, ε, πρέπει να πω ότι αν βρούμε έναν τρόπο να συνεχίσουμε να ε, πιέζουμε την, ε, μέσω της κοινωνίας των πολιτών, μέσω των πολιτών της κυβερνήσης και την Κομισιόν, αυτό θα είναι καλό. Απλώς δεν ξέρω πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Οπότε ας το αφήσουμε έτσι εκρεμές αυτό, ανοιχτό, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για το πώς θα δουλέψει. Ε, δηλαδή δεν μπορώ να, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι μια προσέγγιση παρόμοια με του διαμεσολαβητή θα είναι χρήσιμη. Αλλά αυτά που λέει η έκθεση ε, ξεπερνά τις απλές σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων. Οπότε ας, ας δούμε τι, πώς θα το δουλέψουμε. Ε, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος, αλλά σας λέω και πάλι ότι θα ήταν αρκετά χρήσιμο να ανοίξει έτσι ο δρόμος προς αυτό. Επίσης κάτι άλλο που τίθεται συχνά είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Μόλις ε, μας είπαν να, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το, ε, το ODA, την επίσημη βοήθεια για την ανάπτυξη, που είναι η ραχοκοκαλιά της, ε, των πολιτικών. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και τα, τα κράτη-μέλη θα α, τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ξέρουμε όμως ότι η, συνεχή, η συνεκτική πολιτική σημαίνει όχι μόνο πολιτικές αποφάσεις, αλλά και ε, ε, στοχοθέτηση των μέσων για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Οπότε όταν μιλούμε για την αναγκαιότητα να καθορίσουμε αυτά τα ε, οικονομικά επίπεδα, το κάνουμε για να έχουμε μια συγκεκριμένη συνεκτική πολιτική να μπορούν να υποβάλλονται εκθέσεις για το κράτος μέλος που θα ξέρει τι πρέπει να κάνει για τις κλιματικές αλλαγές, ας πούμε. Αν πούμε ότι θέλουμε να έχουμε επιπλέον επίσημη βοήθεια για ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα, έχει, θα είναι μόνο αυτή η χρηματοδότησή μα. Αλλά θεωρούμε ότι αν δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό αναγνώρισης υποβολή εκθέσεων, τότε μπορούμε να είμαστε πιο ε, δυνατοί. Και μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα χρήματα που δεν ε, ε, αποδίδονται στην ανάπτυξη, αλλά με έναν τρόπο αναπτυξιακό, έτσι ώστε να, είναι, να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτή την, ε, αυτό το νέο τρόπο εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο σύμβουλο του ε, διαμεσολαβητή για πέντε λεπτά έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Χαιρετίζω εξ ονόματος του διαμεσολαβητή τις προτάσεις που υπάρχουν στην έκθεση και που θεωρούμε ότι είναι χρησιμότατες. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή που μας επέτρεψε να εκπροσωπηθούμε σήμερα εδώ. Το 28 άρθρο της Συνθήκης λέει ότι η εντολή του διαμεσολαβητή είναι να ασχολείται με κακοδιοικήσεις ε, στις διάφορες χώρες, αντιπροσωπείες, γραφεία. Η κακοδιοίκηση, η κακοδιαχείριση είναι ευρία έννοια. Ε, όπως αναγνωρίζει η έκθεση, ε, η, υπάρχουν ε, γενικές ε, αρχές όπως αναλογικότητα ή ε, ικανότητα τήρησης της συνοχής που είναι μια αρχή επίσης της καλής της χρηστής διαχείρισης και η συνοχή σημαίνει ότι θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να σέβονται τις υποχρεώσεις που έδωσαν ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωμένες δια νόμου. Η ανακοίνωση το 2005 για τη συνοχή και την ανάπτυξη αποτελεί ένα παράδειγμα μια τέτοια δέσμευση. Δεν είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να φροντίσει για την συνοχή στην ε, πολιτική τη ανάπτυξη. Αυτό είναι δουλειά των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτό μπορεί να κάνει ο διαμεσολαβητή είναι να ελέγξει αν αυτοί οι θεσμοί πληρούν, ανταποκρίνονται στι ευθύνε του και αν χρειαστεί να του βοηθήσει να βελτιωθούν. Η βοήθεια για βελτίωση των θεσμικών οργάνων ουσιωδή στοιχείο του έργου του διαμεσολαβητή και ένα παράδειγμα ήταν η διαμεσολάβηση στην Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλω επίση να σα πω ότι ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή πρόσφατα προσεκλήθη να ενταχθεί στο δίκτυο ανεξάρτητων μηχανισμών λογοδοσία και ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά όργανα όπω το Συμβουλίο Επιθεώρηση Παγκόσμια Τράπεζα αν χρειαστεί, ε, ασκή κριτική ο διαμεσολαβητής σε περίπτωση κακοδίκησης και αυτό το κάναμε όταν έγινε η ε, ανασκόπηση της ε, πολιτικής που ακολουθήθηκε από την τράπεζα για το τρένο στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Οι πολίτες, οι οργανώσεις, ΜΚΟ με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλουν καταγγελία. Ο διαμεσολαβητής ε, συμφώνησε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να ε, ασκήσει τις αρμοδιότητές του και στην περίπτωση ανθρώπων που δεν ε, έμεναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν επρόκειτο για αναπτυξιακά έργα εκτός Ένωσης. Η πρόταση ε, αναφέρεται στις καταγγελίες ε, που χειρίζεται ο ε, διαμεσολαβητής και στην περίπτωση αυτή μια τέτοια καταγγελία θα μπορούσε να είναι το λογικό επόμενο βήμα. Ευχαριστώ. Και τώρα για πέντε λεπτά η κυρία Λαπαλάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε ε, σχόλια στην έκθεση. Ε, το Concorde είναι η ευρωπαϊκή ε, οργάνωση που εκπροσωπεί πάνω από 600 μήκυο σε όλο τον κόσμο ε, ευχαριστούμε την ε, συγγήτρια Φραντσίσκα Κέλλερ για την έκθεση. Οι συστάσεις στην έκθεσή της είναι έγκυρες ε, αναλύουν ε, τις ε, αντιλήψεις των διαφορετικών εμπλεκομένων και θα πρέπει να προσεχθούν και από τις άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το, την Κομισιόν, το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες αυτές. Τώρα που η συνθήκη της Λισαβόνας ε, ε, ανοίγει το δρόμο για νέες πρακτικές και διαδικασίες ε, ε, ώστε να ε, γίνουν αυτά τα ε, προγράμματα. Εμείς πιστεύουμε στη συνοχή, στην ανάπτυξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι πρέπει να στηρίζεται κυρίως στους υφιστάμενους μηχανισμούς. Και έχω κάποιες σχετικές προτάσεις. Καταρχήν, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποβάλει έκθεση δύο φορές το χρόνο για τις εκθέσεις και η Επιτροπή Ανάπτυξης συντονίζει με τη συμβολή των άλλων επιτροπών. Δεύτερον, χαιρετίζομαι την προσπάθεια της εισηγήτριας να προβλέψει διαδικασία υποβολής καταγγελιών αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του οποίου η εντολή θα του ε, της επιτρέπει να ασχολείται με θέματα ε, κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης ή καταγγελίες ε, εκτός που προέρχονται από άλλες χώρες και κοινωνίες των πολιτών εκτός Ένωσης. Τέλος, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει όλες τις επιλογές που έχει, ούτως ώστε οι χώρες εταίροι να συμμετέχουν περισσότερο. Οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να επισκέπτονται τις περιοχές και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις Eurolat, Euromed, ούτως ώστε να ε, γράφονται τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Επίσης ε, ε, εμένομαι στη σημασία των ε, δικτών ανάπτυξης ούτως ώστε να υπάρχει διαφανή συζήτηση για τους δείκτες αυτού αυτούς που θα πρέπει να καταλήγουν σε σημαντικά πρότυπα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ε, πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να αναθεωρούνται αυτές οι πολιτικές αν χρειάζεται και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την, τους δείκτες αηφόρου ανάπτυξης, ε, δείκτες στόχων χιλιετίας κλπ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα εντοπίζουν ε, αστοχίες, έλλειψη συνοχής ε, και μετά θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση των πολιτικών. Θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών στις χώρες να συμμετέχουν πιο πολύ στην ε, ε, κατάρτιση των εθνικών εγγράφων των χωρών, στις διαβουλεύσεις, στις αντιπροσωπίες και η συμβολή τους πρέπει να τεκμηριώνεται ούτως ώστε να υπάρχει απολογισμός των πολιτικών που θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με τη συνοχή ή έλλειψη της συνοχής ανάλογα με τον αντίκτυπο που έχει σε κάθε χώρα. Κυρία Πρόεδρε, υπογραμμίζω ότι η οργάνωσή μας Concord θα θέλει να συμβάλλει αναλαμβάνοντας το ρόλο και την υπευθυνότητά της σε ό,τι αφορά την γενική παρακολούθηση, την αρχιοθέτηση, την προώθηση καταγγελιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις αρμόδιες επιτροπές αναφορών και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Το Κόγκορτ επίσης ε, κατανοεί τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις ε, και ευθύνες ε, προς τους εταίρους και τις κοινωνίες των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, θα ρίνομαι την, τον εντοπισμό πιο έγκαιρα των περιπτώσεων έλλειψης συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ο πρώτος είναι ο κύριος Αρσένης. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Υπογραμμίζει τα διαφορετικά προβλήματα της στρατηγικής. Συμφωνώ και με την ανάγκη μεγαλύτερη εμπλοκή του για μεσολαβητή και του Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι έχει δίκιο όταν ζητά σαφέστερα ορόσημα και δυνατότητες με καλύτερης μέτρησης της πρόοδου. Και είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα, σαφέστερη εικόνα των, της απόδοσης της ανάπτυξης. Συμφωνώ επίσης σχετικά με τις ε, ανησυχίες της για την προσέγγιση αυτή επίσημη ε, ε, ενίσχυση της ανάπτυξης ΣΥΝ και την διεύρυνση ούτως ώστε να περιλαμβούν και άλλες διαστάσεις όπως την ε, χρηματοδοτική ροή κλπ. Επίσης συμφωνώ ότι συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας να υπάρξει συνέχιση της παρακολούθησης των 12 παραδοσιακών τομέων πολιτικής αλλά και των άλλων που θα προτείνει το Συμβούλιο που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συμπληρωματικά. Να προτείνω επίση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη συνέργειας μεταξύ αλλαγή κλίματος και ε, αναπτυξιακών πολιτικών. Ξέρουμε ότι το Ταμείο η χρηματοδότηση προσαρμογής θα πρέπει να έρθει ω συμπληρωματική. Αλλά ξέρουμε τι συνέπειε μπορεί να έχει όταν οι προσπάθειες ε, μετριασμού των, της του κλίματος δεν λαμβάνουν υπόψη την ε, αναπτυξιακή διάσταση και κυρίως τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των χωρών. Κάποιες, ε, κάποια έργα μετριασμού της φτώχειας μπορεί να βελτιωθούν και με, την, με τις πολιτικές αλλαγής του κλίματος. Και αυτό ότι αυτή τη διάσταση δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ κάτι. Ε, ε, ο εισηγητής από τη σοσιαλιστική ομάδα Πατρίς Ρουλέν δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Καταρχήν να συγχαρώ τη Φραντσίσκα Κέλλερ για λογαριασμό του. Είναι εξαιρετική έκθεση που μας επιτρέπει να κάνουμε καλή συζήτηση σήμερα. Φαίνεται ότι βελτιώσεις μπόρεσαν να γίνουν στο σχέδιο έκθεσης μετά από τις παρατηρήσεις μας. Θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη τομεακών πολιτικών της Ένωσης, όπως εμπόριο, γεωργία, αλληλεία, για παράδειγμα, που δεν ε, αναδεικνύονται τόσο πολύ, δεν αναδεικνύονταν στο σχέδιο έκθεσης. Γι' αυτό κάναμε και κάποιες ε, τροπολογίες για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής που βάσει συνθήκες Λισαβόνας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτικές, εξωτερικές και εσωτερικές, ώστε να πληρούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι της Ένωσης. Η Κομισιόν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ε, ΣΑΠ, Συνοχή Αναπτυξιακής Πολιτικής, ε, θα πρέπει να ε, βελτιώνει και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη. Ο ορισμός αυτής της ε, έννοιας είναι ασαφής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ε, αντίκτυπο που έχει στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Πάνω στη βάση αυτής της ολιστικής προσέγγισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε πέντε τομείς προτεραιοτήτων σε αντιπαράθεση με 12 που ήταν πριν η ΣΑΠ. Επίσης, το Συμβουλίο ασχολήθηκε με τις προτάσεις της Κομισιόν συμπεριλαμβάνοντας εμπόριο και ε, ε, χρηματοπιστωτικό δημοσιονομικό τομέα. Ε, έτσι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περισσότερο η ε, ανησυχία και τα προβλήματα των αναπτυσσευμένων χωρών. Η Κομισιόν προτείνει επίσης ε, να εντοπίσουμε και να προαγάγουμε τις ε, μη χρηματικές ροές προς τις χώρες που αναπτύσσουν την νέα αυτή αντίληψη περί επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας ΣΥΝ. Ορίζεται η ΕΑΒ, Αναπτυξιακή Επίσημη Βοήθεια, με αξιέπαινη συνέπεια. Δεν γίνεται αναφορά ε, εις ό,τι αφορά κάποια δισεκατομμύρια ροές από τον νότο προς το βορρά που έχουν τελείως διαφύγει ε, από το κείμενο και από τις φορολογικές αρχές ε, των βορείων χωρών. Θα πρέπει όμως και ο Βορράς και ο Νότος να συνεργαστούν στη διαταπολέμηση της φτώχειας και ε, ε, στην προαγωγή της ενότητας, της ε, ισότητας. Θέλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε ούτω ώστε να υπάρξει περισσότερη συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στη δημοσιονομική διαχείριση. κυρία Σνάιμπερ Σέντραμ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Φραντσίσκα Κέλλερ για την ωραία έκθεση. Ευχαριστώ επίσης και για τις καλές συζητήσει που προηγήθηκαν του σχεδίου έκθεσης, γιατί συμφωνήσαμε εν πωλής και επί του περιεχομένου της έκθεσης. Ε, έχω μερικά πράγματα όμως που θέλω εν συντομία να παρατηρήσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα δυνατότητα να ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπο του διαμεσολαβητή κάποια πράγματα, γιατί το θέμα αυτό είναι ευρύτατο. Και το ερώτημα αν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο ο διαμεσολαβητής ε, με τα μέσα που διαθέτει, το έχει απαντήσει ήδη θετικά. Έχω κάποιες ελαφρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να τα καταφέρει ακούγοντας ε, το πώς οι συνεργάτες αυτής της Επιτροπής ε, παραπονούνται πολλές φορές για την ε, υπερβολική εργασία, το μεγάλο φόρτο εργασίας. Και πού μπορεί, ποιος μπορεί να ε, υποβάλει μια καταγγελία, ο Πάσα ή μόνο τα θεσμικά όργανα και τι συνέχεια δίνεται στις καταγγελίες που υποβάλλονται και πώς μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Αυτά Νομίζω ότι είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί ο στόχος μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Προφανώς θέλουμε ισχνούς θεσμούς που να μπορούν να λειτουργούν και να επισημαίνουν τα σφάλματα. Πού δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες αναπτυξιακές σε άλλους τομείς που δεν ελήφθησαν υπόψη. Το βασικό ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε αυτό το στόχο που έχει θέσει η Φραντσίσκα Κέλλερ, να υπάρχει κάποιος συνομιλητής ο οποίος ε, να μπορεί να παρεμβαίνει και να χειρίζεται τα θέματα. Είναι δύσκολο ο τομέας νομίζω. Ε, μπορούμε βέβαια και με τροπολογίες να δουλέψουμε εδώ και να προσθέσουμε για παράδειγμα ότι το εμπόριο σε αυτούς τους τομείς της πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνεται. Το Συμβούλιο ήδη νομίζω το έχει συμπεριλάβει αυτό, το έχει δεχτεί και μπορούμε να το ρυθμίσουμε μέσα από τροπολογίες. Αλλιώς υπάρχει μεγάλη συμφωνία με την έκθεση αυτή και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ στην εισηγήτρια. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με τα συγχαρητήρια προς την κυρία Κέλλερ για την έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή καλύπτει δύο βασικά θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής. Πρώτον, την συνέπεια των πολιτικών αυτών. Για πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοζε την βιβλική αρχή μη γνώτο η αριστερά, τύπη η δεξιά. Κάτι εξαιρετικά κακό όταν θέλουμε να λύνουμε προβλήματα, γιατί όλες οι πολιτικές της Ένωσης και το αριστερό και το δεξί χέρι πρέπει να δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλιώ ό,τι προσπαθούμε να πετύχουμε με το ένα χέρι το γκρεμίζουμε με το άλλο κατά πάση Πιστεύω ότι μπορεί να δοθεί μια κάποια ευελιξία στους τομείς συνοχής, όχι όμως τόση όση αυτή που εφάρμοσε η Επιτροπή και που υπογραμμίζει στην έκθεσή της η κυρία Κέλλερ. Δηλαδή, ε, υπάρχουν τομείς όπως ε, η χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση ή η ενέργεια που αυτή τη στιγμή σε εποχές οικονομικής και ενεργειακής κρίσης είναι βασικές παράμετροι για να εξετάσουμε τις πολιτικές ανάπτυξης. Το δεύτερο μεγάλο θέμα αφορά στην, αναπτυξη, στην συμπληρωματική αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύω ότι παρότι η Επιτροπή ε, έδειξε, είχε επιφυλάξει προς το αν θα κρατήσει το ζήτημα αυτό στο μέλλον ή όχι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε προσεκτικότερα. Όχι σήμερα κατά ανάγκη, αλλά κάποια στιγμή, διότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι συγκεκριμένες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές ε, ροέ που καθοδηγούν την αναπτυξιακή βοήθεια να συνυπολογίζονται σαν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, έτσι για να μπορέσουν τεχνητά να πούν οι χώρε ότι τήρησαν τι δεσμεύσει του και αποδυναμώνοντα την πραγματική αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Πιστεύω ωστόσο ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα κλειστοί και αρνητικοί στον συμπολογισμό νέων έκτακτων μορφών χρηματοδότησης ζητημένου στόχους, προκαθορισμένους, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ε, υφιστάμενες αναπτυξιακές πολιτικές. Δηλαδή, αν υπάρχουν χώρε που θέλουν να συμβάλλουν συμπληρωματικά σε σαφώ αναπτυξιακά, ξεκάθαρα αναπτυξιακά έργα, που δεν είναι αυτά που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα πρέπει να ε, απογοητεύσουμε τι χώρε αυτέ λέγοντα ότι τούτο δεν θα συμπεριληφθεί στην, στον υπολογισμό τη συνεισφορά σα για την ανάπτυξη. Δεύτερο, και τελειώνω, η έκθεση θα μπορούσε να δώσει λίγο περισσότερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Κάτι που θεωρούμε σημαντικό για να χτυπήσουμε την ε, ασυνέπεια. Να πω και κάτι ακόμα. Συμφωνώ με κάποιες προηγούμενες παρεμβάσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι το θεσμικό σχήμα που παρουσιάζει η πρόταση είναι υποχρεωτική με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εγώ θα έλεγα γιατί είμαι κάπω ετερόδοξο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει, ότι είναι πιο σημαντικό να υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ των βασικών οργάνων της Ένωσης, Επιτροπής Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, από ότι να περάσουμε ε, κάποια στοιχεία στις καταγγελίες σε ένα όργανο που αφορά παράπονα πολιτών. Προφανώς η καταγγελίες για ασυνέπειες στην πολιτική ανάπτυξη θα πρέπει να απευθύνονται και που απευθύνονται και συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι πιο χρήσιμο να δουλεύει από κοινού Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την τήρηση των πολιτικών συνοχής. Αυτά και συγχαρητήρια εκ νέου στην εισηγήτρια. Καλή επιτυχία για την έκθεσή σας. Θα προσπαθήσουμε να την βελτιώσουμε σε πολύ λίγα σημεία με κάποια μικρή τροποποίηση. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο σε όλους τους ε, αγωγητές. Ο κ. Μανσερβίση για την Επιτροπή. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σύντομα. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις έδειξαν τη σημασία και τον κεντρικό χαρακτήρα του θέματος για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί πληρέστατα με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτή η ημερήσια διάταξη. Συνεχίζω να πιστεύω έστω και ότι ε, διαφωνείτε ότι εμείς δεν μιλάμε για ODA συν, ΕΑΠ εγώ, αλλά ε, οι πράξεις θα δείξουν. Συμφωνώ με πολλοί με αυτά που είπε ο κύριος Γεραίρο. Πρέπει να δώσουμε στο εργαλείο συνοχής κάποια περισσότερα, κάποιες περισσότερες δυνατότητες. Να καταλάβουμε κάτι, τα άλλα πράγματα που κάνουν για την ανάπτυξη στα κράτη, χωρίς να χρειαστεί να ε, παρεκφύγουν ή να καταστατηγήσουν τη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας. Λέω λοιπόν, δεν μιλάμε για εαψίν, εαψίν αλλά για κάτι συμπληρωματικό. Τρίτο θέμα. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Το θέμα δεν είναι ένα θέμα ε, που δεν αφορά εσάς. Προφανώς γι' αυτό ε, υπάρχει και ο διαμεσολαβητής. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε με, με κάποια ορόσημα τι θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατηφόρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής που έκαναν παρατηρήσεις για τον διαμεσολαβητή. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Σράιμπερ που αυτή τη στιγμή νομίζω δεν είναι εδώ. Ο, Ευ... Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δέχεται 3 με 4 χιλιάδες καταγγελίες ετησίως από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μη κυβερνητικέ οργανώσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Τώρα, η παραλαβή ε, καταγγελιών σε σχέση με το ε, θέμα μας και το αν αυτό θα επιβάρυνε υπερβολικά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά αυτό το είναι θέμα αριθμού βέβαια, πόσες καταγγελίες θα ε, υποβάλλονταν γι' αυτό. Ένα παράδειγμα, έχουμε ένα ε, μνημόνιο συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το τις δραστηριότητε της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή βάζοντας καταγγελίες και από υπηκόους τρίτων χωρών. Μέχρι τώρα αυτό ε, το συνήψαμε, το, μνημόνιο, πριν από 18 μήνες και δεν είχαμε ακόμα ούτε μία καταγγελία στα πλαίσια αυτού του μνημονίου συνεννόησης. Τώρα, ποιος μπορεί να υποβάλει μία καταγγελία. Αν η καταγγελία απευθύνεται κατά κοινοτικού θεσμού ή ε, οργανισμού οποιοδήποτε μπορεί να καταγγείλει ακόμα και αν είναι υπήκος τρίτης χώρας και ο Ευρωπαίος Διάμεσολαβητής θα πρέπει να ασκήσει ε, τις εξουσίες του πρωτοβουλίας για να δεχτεί την καταγγελία. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα σχόλια που ακούστηκαν από όλους. Όντως υπάρχει μεγάλη ε, ε, εμπλοκή της ε, Επιτροπής σας για το θέμα αυτό και βεβαίως καλωσορίζουμε τα σχολεία σας. Είναι σημαντικό για μας αυτές οι συζητήσεις να συνεχίσουν. Εμείς θα υποβάλουμε την έκθεσή μας, υποβάλαμε μάλλον την έκθεσή μας ήδη από το φθινόπωρο με συγκεκριμένες περιπτώσεις για εμπόριο, μετανάστευση, ασφάλεια, οικονομικά κτλ για να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώ αυτέ τι αποδείξει για την ε, συνοχή στην πολιτική και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με δεδομένο και τα παραδείγματα που έχουμε αλλά και ε, με τη δική σα βοήθεια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε του ε, δείκτε για την καλύτερη συνοχή για την αναπτυξιακή βοήθεια και ακόμη πρέπει να βρούμε τον σωστό μηχανισμό υποβολή παραπώνων για να δούμε πώ μπορούμε να καταδεικνύουμε τι αποδείξει όταν υπάρχουν ασυνέπειε και κακοδιαχειρήσει. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα αυτό και βεβαίω αν χρειαστεί μπορούμε να επανέλθουμε εδώ ενώπιόν σα για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο κυρία Κέλλερ για τα καταληκτικά σας σχόλια. Λίγα λεπτά. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη και την συνεισφορά που παρουσιάζετε, τις συνεισφορές που παρουσιάζετε. Θα, δεχθώ, θα εξετάσω ευνοϊκά τις παρατηρήσεις, ιδίως τις προσφύγκες, για παραδείγματα κλπ. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες προσθήκη. Περιμένω λοιπόν τροπολογίες. Εγώ γιατί σκέφτηκα ότι καλή ιδέα είναι ο διαμεσολαβητής, γιατί υπάρχει. Είναι το γραφείο του διαμεσολαβητή, δεν χρειάζεται να υπάρξουν νέα γραφεία που θα πάρουν δύο χρόνια. Ε, έχει την εμπειρία. Μας είπατε ίσως ότι έχει ε, ήδη μεγάλη εμπειρία από καταγγελίες για κοινοτικά όργανα και αφορά ακριβώς ε, ασυνέπειες συμπεριφορών των κρατών μελών. Γι' αυτό είπα να ο διαμεσολαβητής, γιατί υπάρχει, να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτά, ευχαριστώ και ελπίζω να λάβουμε περισσότερα στοιχεία και προτάσεις για να βελτιωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την, για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 12 η ώρα το μεσημέρι στις 4 Μαρτίου. Τώρα θα μπούμε στο επόμενο σημείο δια... της σημερινής στην την στρατηγική της Ένωσης για τη σχέση με τη Λατινική Αμερική. Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Δεν το βρίσκεται στο ντοσχέ σα. Διανεμήθηκαν οι εκδοχές στα αγγλικά και τα γαλλικά. Αν χρειάζεστε άλλη γλώσσα, ζητήστε το κείμενο από τους ε, κλητήρες. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να δώσω το λόγο αμέσως στη συνάδελφο κυρία Γκρέζ για να μας παρουσιάσει τα βασικά θέματα του κειμένου. Πέντε λεπτά έχετε το λόγο κυρία Γκρέζ. Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε τεχνικό πρόβλημα. Ομολογώ πως είναι πολύ δύσκολο να δουλεύουμε κάτω από τις συνθήκες αυτές. Πριν από 13 μέρες έδωσα την έκθεση όταν μου το είχατε πει. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν σε μια μισή μέρα. Αλλά μετάφραση γιοκ. Οι συνάδελφοι τώρα φαντάζομαι ότι βλέπουν το κείμενο. Τέλος πάντων, τάπα να επανέλθω τώρα στο βασικό θέμα και να υπενθυμίσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής 16-17 Μαΐου στη Μαδρίτη. Ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής είναι ο ρόλος της καινοτομία και της ε, τεχνολογίας σαν εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης. Η Επιτροπή Εξωτερικών βέβαια είναι αυτή που αποφασίζει επί της εκθέσεως, αλλά προφανώς η δική μας Επιτροπή ενδιαφέρεται από, για θέματα όπως τη μάχη κατά της φτώχειας, τους στόχους της ηλικίας και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και άλλωστε από το ξεκίνημά μας οι εργασίες μας προσβλέπουν σε, μια, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που έχει ως προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή, το σεβασμό των δικαιωμάτων ανθρώπου και του περιβάλλοντος τα κείμενα που μας υποβλήθηκαν και οι εργασίες επιτροπής δείχνουν ότι οι προτεραιότητες της Ένωσης εστιάζονται κατά βάση στις εμπορικές συνταλλαγές με την Λατινική Αμερική και μόνο, και υπογραμμίζω το μόνο, δευτερευόντως σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της φτώχειας και πιστώνουμε ότι η πολιτική διάσταση και η διάσταση δικαιών του ανθρώπου χάνουν ε, την σπουδαιότητα ενώ ενώπιον των εμπορικών ε, διαπραγματεύσεων. Μέσα στο πλαίσιο τη μεγαλύτερη κρίση σήμερα για την Λατινική Αμερική από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80, που δείχνει ότι οι πολιτικέ που επιβάλαμε δεν καρποφόρησαν, επιπλέον έχουμε και παράλληλα την αποτυχία τη Κοπενχάγη με μια μελέτη που δείχνει ότι η Λατινική Αμερική ε, πλήττεται ιδιαίτερα από την αλλαγή του κλίματο και ότι μέχρι το 2100 το 40% της βιοπικιλότητας στην υποήπειρο θα εξαφανιστεί. Διαπιστώνουμε ταυτόχρονα ότι οι λύσεις που, θέτουν, ε, που προτείνουν οι πλούσιες χώρες για τη δημιουργία μηχανισμών αυτόνομης ανάπτυξης δεν είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικ τοπική πραγματικότητα και συχνά παραβιάζουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Για να βγουν λοιπόν από την κρίση οι χώρε τη Λατινική Αμερική, πιστεύουμε ότι οι λύσει θα πρέπει να στηρίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση τη κοινωνική κατάσταση και τη περιβαλλοντική κατάσταση τη Υπήρου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνει την προτεραιότητα των σχέσεών της αυτών με τη Λατινική Αμερική, να κάνει όπως προτεραιότητα τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος και τη μάχη κατά της φτώχειας. Η, η Ένωση θα πρέπει να προσβλέψει στη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων για το περιβάλλον και στη μάχη κατά της φτώχειας. Δεν πρέπει να είναι απλά εμπορική η προσέγγιση αυτή. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργηθεί μια πραγματική σχέση και να αποφευθεί η συμφωνία που δεν θα τηρεί τις προϋποθέσεις αυτής, ενώ θα συμβάλλει στην, ε, στον κατακαιρματισμό της κοινότητας των άνδρων. τι προάλλες είδαμε πώς, ε, πόσο κακό παράδειγμα είναι οι διαπραγματεύσεις ε, που διεξάγονται με Περού και Κολομβία. Ζητούμε λοιπόν μεγαλύτερο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καταπολέμηση κατά τη φτώχεια, καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος και δέσμευση ότι όλε οι συμφωνίε Ευρώπης και Λατινική Αμερική θα λαμβάνουν υπόψη αυτές, αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. La parole est au député. Οι κύριοι και οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης υπογραμμίζει ιδίω τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δικαίω, διότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η πρώτη γραμμή, μια γραμμή που δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί. Για την αντιμετώπιση ωστόσο της κρίσης στη Λατινική Αμερική χρειάζεται και κάτι παραπέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε η γνωμοδότηση να ασχοληθεί με μια σειρά θεμάτων που θα ασχολούνται με τον παγκόσμιο σφαιρικό στρατηγικό χαρακτήρα που έχει το σύνολο των σχέσεων της Ένωσης με τη Λενική Αμερική. Να σας πω κάποια θέματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν κατά την άποψή μου στο σχέδιο γνωμοδότησης και που θα στείλω ως ε, τροπολογίες ή θα θέσω στην εισηγήτρια πάντων για να τις λάβει υπόψη της εάν συμφωνεί. Πρόκειται για στα εξή θέματα. Να φέρουμε τη δυνατότητα να δρούμε από κοινού, η Λατινική Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις ε, υφιστάμενες διαδικασίες ε, σφαιρικού χαρακτήρα στον κόσμο. Τη μεταρρύθμιση των ε, οικονομικών φορέων, θα συνεχίσει σε λίγο το G20, την αλλαγή του κλίματος. Δεν είναι τυχαίο το ότι στο Μεξικό θα πρέπει να ληφθεί μια τελική απόφαση για την αλλαγή του κλίματος και την τήρηση των στόχων της Χιλίτιας. Εάν πάρουμε μαζί τις χώρες της Ένωσης και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, βλέπουμε ότι είμαστε ένα ουσιαστικό, σημαντικό κομμάτι του συστήματος του ΟΗΕ, της παγκόσμιας παραγωγής και, της και του παγκόσμιου πληθυσμού. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο κάτοικοι. Είναι η στιγμή λοιπόν για αυτά τα παγκοσμιοποιημένα πλαίσια που ανέφερα, μέτρα κατά της κρίσης, αλλαγή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλαγή του κλίματος, στόχοι της χιλιαστίας, πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού εν ώψη της, ε, Συνόδου της Μαδρίτης που θα γίνει το Μάιο για να πετύχουμε κοινέ θέσεις που θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στους διάφορους πολυεθνικούς φορείς. Να σας πω ότι συμφωνώ με βασικά κομμάτια της γνωμοδότησης την ανάγκη διαφάνειας φορολογικού χαρακτήρα, την, το σεβασμό των αυτοχθόνων, την πρόσβαση στις ε, δημόσιες υπηρεσίες, όπου θα συμπεριλάμβανα και το θέμα της υγείας, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα στη Λατινική και Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εν γέννη συμφωνώ με τις ιδέες ε, που παρουσιάζει η κυρία Γκρέες. Συμφωνούσα και με τη δράση του συζύγου της Didier κατά τη διάρκεια των περασμένων 10 ετών όταν συνεργαζόμασταν δίπλα-δίπλα και με την ευκαιρία να του στείλω την αγάπη μου. Να πω και κάποια πράγματα για αυτά που είπε και η κυρία Γκρέζ και ο συνάδελφος κύριος Γκερέρο. Με εξέπληξαν κάποια από αυτά που είπε η κυρία Γκρέζ, γιατί δεν τα βλέπω στο κείμενο. Δεν βλέπω να υπάρχει επαρκή έμφαση στο θέμα της μάχης κατά της φτώχειας, στο θέμα της μάχης για την επίτευξη των στόχων, των απτυξιακών στόχων της χιλιεστίας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να μετέχουν, να είναι κομμάτι, στο κείμενο που θα στείλουμε εμείς στην Επιτροπή Εξωτερικών. Δεν έχω λίγα ε, συγκεκριμένα σχόλια, λίγα μόνο. Θεωρώ πολύ σημαντικό όταν λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσπισή τους αποτελούν λύση για την κρίση. Για την κρίση καλύτερα θέλετε να πούμε ότι είναι τμήμα της λύσης για την κρίση. Υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαντικά στοιχεία. Όταν μιλάμε τώρα για πολιτισμικά δικαιώματα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κοινωνικοπολιτισμικά δικαιώματα. Γιατί μιλάμε, ε, μιλάμε για πολιτικά, για, για ανθρώπινα, για περιβαλλοντικά δικαιώματα ε, και για πολιτισμικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να αγνοήσουμε τα κοινωνικο-οικονομικά. Α, κάτι ακόμα. Μια μέρα, σαν τη σημερινή, που σε πολλές χώρες ε, ε, είναι η μέρα της καταπολέμησης των διακρίσεων κατά των γυναικών ιδιότητες ό,τι αφορά το μισθολογικό χαρακτήρα. Έχω την εντύπωση ότι κάπως ανακατεύουμε τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των αυτόχθονων, που δεν είναι σωστό. Με άλλα, δηλαδή, ε, υπάρχουν γυναίκες αυτόχθονες που υφίστανται ε, διάκριση και ως γυναίκες και ως κομμάτι αυτόχθονων πληθυσμών. Κάτι άλλο. Όσοι με ξέρετε, το λέω, ξέρετε, το λέω και το ξαναλέω. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να υποστηρίζει την, ε, την εξομάλυνση των σχέσεων της Ένωσης με την Χούβα. Είναι κάτι που σε πολλές χώρες ε, τίθεται. Το ζήτησαν όλες οι χώρες της Ελληνικής Αμερικής, το ζητούν οι χώρες ΑΚΕ συστηματικά. Πιστεύω ότι και εμείς μέσα στη γενική παρέμβασή μας για, τη, ε, ε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουμε την, την, ε, ε, την Κούβα, αλλά δεν μπορεί να περιορίζουμε μια χώρα. Θα πρέπει να προβλέπουμε ότι να ζητούμε μια εξομάλυνση των σχέσεων μέσα στο πλαίσιο, το ευρύτερο πλαίσιο της έκθεσης της κυρίας Γκρέζ. Ευχαριστώ. La Κύριος Thank you very much. Ε, would like to... Ευχαριστώ. Να συγχαρώ την ησυχήτρια γιατί επικεντρώνεται και στο κλιματική αλλαγή και στα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών για την ε, κλιματική αλλαγή. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά για την ε, Λατινική Αμερική, είναι το θέμα του νερού και το ε, λιωσίματος των παγετώνων. Πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με λήψη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Οπότε ίσως θα πρέπει κάτι να αναφέρετε στην εκθέσή σας από αυτού. Και για την κλιματική αλλαγή και πάλι, για τα δάση. Υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την φυσική αναδάσωση. Γιατί τώρα το βασικό πρόβλημα είναι η αποψήλωση. και επίσης για τις σεξουαλικές ε, βιομηχανίες, οι οποίες επίσης απειλούν τα δικαιώματα των ε, αυτοχθόνων. Το έχουμε πει πολλές φορές και οι δυστυχώς οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείες, επιχειρήσεις συμβάλλουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρεντς, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέζ για το κείμενο που μας παρουσίασε. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Σημείο 3 που αναφέρεται οικολογική, το οικολογικό χρέος της Ένωσης προς τις χώρες ε, της, της ε, Λατινικής Αμερικής. Υποτίθεται ότι μιλά, φαντάζομαι ότι μιλά για τους, ε, τις ευθύνες για τις οποίες θεωρεί η κυρία Γκρέσου ότι η Ένωση είναι υπεύθυνη. θα ήθελα να ακούσω κάτι περισσότερο γι' αυτό. δεν νομίζω ότι είναι ένα επίσημο θέμα που μπορούμε να το θέσουμε σε διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, δεν, έχω καταλάβει. Θα ήθελα κάποιες περισσότερες εξηγήσει. Κατόπιν. Σημείο 5. Ζητείται η αναγνώριση της επισητιστικής κυριαρχίας. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο επισητιστική ασφάλεια και όχι επισητιστική κυριαρχία. μπορούμε να το δούμε σε εθνικό επίπεδο αυτό να, ή σε περιφερειακό αλλά αυτό δεν, αν το δούμε περιφερειακά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κυριαρχία κάθε χώρας ε, μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς ε, επιστημιστική ασφάλεια χωρίς να έχει επιστημιστική κυριαρχία πάντα και σε όλα. Κάτι άλλο. Μιλάει η κυρία Γκρέ για τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις. Εγώ θα έλεγα η διατύπωσή της να είναι λίγο πιο θετική για τις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτά. Και να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Γκρέζ. Δεν μπορώ να στείλω χαιρετίσματα στον άντρα της, γιατί δεν τον ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Ο κύριος Μπέζ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρές για τα σχόλιά της στην έκθεση του κυρίου Σαλαφράγκα που ήδη είχαμε καλωσορίσει όταν είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επιτρέψτε μου κάποια σχόλια που αναδεικνύουν την παρουσίαση, καταρχήν τα θέματα φτώχειας που αναφέρονται στο κείμενο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάνω από το 40% της συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική αφορά τη κοινωνική συνοχή και ασχολούμεθα με κάποια θέματα που αναφέρονται και εδώ. Για την κλιματική αλλαγή που ανέκυψε επίσης η αλλαγή του κλίματος αναφέρεται με τρόπο οριζόντιο σε όλα τα έγγραφα που λαμβάνει το Κοινοβούλιο ε, ή θα λάβει. Είναι προτεραιότητα και θα συνεχίσει να είναι. Στα πλαίσια του περιφερειακού εγγράμμου στρατηγικής έχουμε αναφορά στο κλίμα που ασχολείται με αυτά τα θέματα σε περιφερειακό επίπεδο στην Λατινική Αμερική. Και το, η επενδυτική ευκόλυνση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη εδώ. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε σε συνεχή διάλογο με την περιοχή αυτή και ε, κάνουμε ειδικού διαλόγους με κάποιες χώρες ε, και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό και 20% των ε, παρεμβάσεων σε πλαίσια αυτού του προγράμματος πάνε στη Λατινική Αμερική. Τέλος, για τη Συμφωνία Σύνδεσης, όπως ξέρετε η Κομισιόν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες αυτές τις ημέρες στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων συμφωνιών σύνδεσης με διάφορες υποπεριφέρειες της Λατινικής Αμερικής και γνωρίζετε ίσως ότι δεν είναι μόνο εμπορικά θέματα που συζητούνται εδώ, που τα διαπραγματευόμαστε. Ο στόχος είναι στο τέλος να υπάρχουν συνολικές συμφωνίες που θα άπτονται και πολιτικών, και οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το θυμόμαστε. Σταματώ εδώ και σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκρέσ, εντάχει για να κλείσετε, παρακαλώ. Τώρα μην, ε, ούτως ή άλλως έχω να κάνω και μια άλλη έκθεση, μια άλλη επιτροπή σε 10 λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους, τους ομιλητές για τα πλούσια, ε, για τις πλούσιες παρεμβάσεις τους, για τις παρατηρήσεις που έγιναν για τις γυναίκες και τους αυτόχθονες λαούς. Αλλά και για το σημείο 7 στη διατύπωση που λέει ότι πρέπει να είναι θετική επίσης την ανοιχτή σε ό,τι αφορά την ανάγκη διατήρησης της κοινότητας των άνδρων. Τώρα για το θέμα επισυντιστική ασφάλεια, επισυντιστική κυριαρχία, νόμιζα ότι το είχαμε συζητήσει και το είχαμε κλείσει στο παρελθόν σε μια έκθεση του κυρίου Μαρτίνες εδώ, όταν ο όρος κυρι... είχε... όπου είχαμε προτιμήσει τον όρο επισυντιστική κυριαρχία. Τέλος πάντων θα εξετάσω την πρότασή σας. Κατέγραψα τα σημεία που αναφέρατε και τα νέα στοιχεία για την εξομάλυση των σχέσεων Ένωση Κούβα. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σα ζητούσα πάντω την επόμενη μία μισή μέρα να προσπαθήσετε να με βρείτε για να ετοιμάσουμε ένα κείμενο τροπολογιών από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Προθεσμία κατάθεσης απολογιών 26 Φεβρουαρίου μεσημέρι. Προπολογισμό. Εντάχει. Κα, κατευθυντήριε γραμμέ. Η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Προλογισμών, ψηφίζει στι 4 Μαρτίου τον προπολογισμό. Θεωρήσαμε σκόπιμο η Επιτροπή μα να μπορέσει να πει κάτι για τον επόμενο προπολογισμό ήδη στη φάση αυτή τη διαδικασία. Όμως επειδή υπάρχει πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ε, πρέπει να βιαστούμε αν θέλουμε να έχουμε μία γνωμοδότηση. Λοιπόν, τα σχέδια γνωμοδότηση υπάρχουν στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ο εισηγητής είναι ο κ. Μπέρμαν. Χρειάστηκε να πάει στην Ολλανδία γιατί έχει, μια, έχει κρίση κυβέρνηση εκεί, έπεσε κυβέρνηση όπως ξέρετε. Μου έδωσε τι ήθελε να σας πει το σημείωμά του. Σας το διαβάσω. σας τονίζω ότι η προθεσμία των υπολογιών είναι Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, μεσημέρι, 12 η ώρα, στα αγγλικά. Φέτος πήραμε την δεύτερη ενδιάμεση έκθεση για τους στόχους της χιλιετίας που είναι η, ο στόχος για την επίτευξη του στόχου ενίσχυ, βοήθεια 0,56%. Αυτό δεν ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη. Με αυτό το σκοτεινό πλαίσιο και, την, και το υφιστάμενο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης φοβούμε ότι ε, η κατηγορία 4 πραγματικά είναι πολύ τραβηγμένη. Κατά την άποψή μου, θα κάνουμε, προτείνω να κάνουμε τέσσερις, κάποιες ε, προτάσεις στην Επιτροπή Υπολογισμών που θα επιτρέψουν την Επιτροπή να μειώσει το, τα προβλήματα που οι περισσότερε φτωχέ χώρε αντιμετωπίζουν. Αλλαγή κλίματο. Η αλλαγή του κλίματο δημιουργήθηκε από τα βιομηχανικά κράτη, ενώ το τίμημα το πληρώνει οι φτωχέ χώρε. Εκτιμάται ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε αντιμετωπίζουν 100 δις ευρώ το χρόνο δολάρια ε, δαπάνε εξαιτία τη αλλαγή του κλίματο. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για το μετριασμό των συνεπειών τη αλλαγή του κλίματο. Μετά την απογοήτευση της Κοπενχάγης χρειαζόμαστε να έχουμε ε, σοβαρή δέσμευση στον προπολογισμό του επομένου έτους για την αλλαγή του κλίματο. Προσβλέπω στην Επιτροπή για να βρούμε το σωστό εργαλείο να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν και να μετριάσουν και να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος. Η οικονομική κρίση. Δεν ήταν αρκετή η αλλαγή του κλίματος. Έπεσε και η οικονομική κρίση η οποία ε, έπληξε τι φτωχέ χώρε εξαιτία των πλούσιων χωρών ή πιο σωστά εξαιτία των ε, παράλογων κερδοσκοπικών ε, συμπεριφορών κάποιων και ε, κλάδων στις πλούσιες χώρες. Τα κράτη και παίρνουν σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κάμψης, αλλά άλλες χώρες εκτός ΑΚΕ δεν το κάνουν. Στον προϋπορισμό του 10 εξασφαλίσαμε μια προπαρασκευαστική δράση για χώρες ε, επίσημης αναπτυξιακής ε, βοήθειας με ένα προϋπορισμό 3 εκατομμυρίων. Υποστηρίζω ε, μια εκθετική αύξηση στη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών για το 2011. Η IT, η οποία όπως ξέρετε επλήγει από τον χειρότερο σεισμό των τελευταίων δύο ετών με πάνω από 200.000 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Η χώρα ε, υφίσταται τώρα μια φρικτή κρίση, όχι μόνο ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και τεράστιες προκλήσεις ανοικοδόμησης. Η, ανταπο, η ανταπόκριση της Ένωσης ήταν γρήγορη και ουσιαστική, ωστόσο ε, υπήρξε, σοβαρό, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού επιτόπου από πλευρά διαφορετική, λόγω διαφορετική συμπεριφορά των ε, δωρητών. Πρέπει να ενισχύσουμε τι προσπάθειε ε, συντονισμού μεταξύ των δωρητών, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων κλπ. Επίσης χρειαζόμαστε κονδύλια για να χρησιμοποιηθεί γρήγορα η ανθρωπιστική βοήθεια. Μικροπιστώσεις και επιστημιστική ασφάλεια. Η κρίση του 2008 στα τρόφιμα έπληξε τους πιο φτωχούς ανθρώπους ε, στον κόσμο. Ε, το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου για την επιστημιστική βοήθεια μόνο ελάχιστα μπορεί να κάνει και πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βοήθεια στους μικρούς γεωργούς, γυναίκες ιδίω να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στα τρόφιμα και την επιστημιστική ασφάλεια. Είναι, ήταν σωστή η προσέγγιση των προϋπολογισμών του 9 και του 10 να υποστηρίξουν προγράμματα μικροπιστώσεων και ζητάμε να συνεχιστούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ζητώ από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον προπολογισμό για να δώσει καλύτερη προτεραιότητα, μεγαλύτερη προτεραιότητα και πρόσβαση στις οικονομικές υπηρεσίες σε αναπτυσσόμενες χώρες και πρόσβαση στις, στην ε, ενίσχυση των ασφαλιών ε, της ασφάλισης των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. σε ό,τι αφορά τώρα το εργαλείο αναπτυξιακή βοήθεια, το εργαλείο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο δημιουργήσει η Επιτροπή ε, πρέπει να έχει επαρκέ προσωπικό και ε, είναι κρίμα το ότι η Επιτροπή έχει αυτή τη στιγμή μικρότερους, ε, μικρότερο, μικρότερο αριθμό εργαζομένων για την αναπτυξιακή βοήθεια από κάποιες ΜΚΟ. Πρέπει να υπάρχουν καινοτόμε μορφέ χρηματοδότηση. Είναι κρίμα το ότι μα υποχρεώνει η Επιτροπή Προπολογισμού να, δι, να δουλεύουμε σε τόσο πιεστικά χρονικά πλαίσια που δείχνει, ή τέλο πάντων μοιάζει να δείχνει ότι θέλει να αποφαρύνει τι άλλε επιτροπέ από το να παρεμβαίνουν. Αυτά. Οι συνάδελφοι έχετε το λόγο. Κύριε Μίτσελ. Πρόεδρε, είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή και Όντως υπάρχει αλλαγή στην χρήση της χρηματοδότησης και θα συμφωνήσω γενικώ με το κεντρικό νόημα της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you. Then the floor is for the Commission. And uh, you don't have any comment? Okay. Um, you have until the 24. th 24 Φεβρουαρίου ε, στις 12 το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και επειδή δεν έχουμε πολύ καιρό μέχρι την Τετάρτη, ε, οι τροπολογίε στα γαλλικά ή στα αγγλικά παρακαλώ, σε όχι, όχι σε άλλες γλώσσε. Τώρα, περιμένουμε τον ε, Επίτροπο. Ε, μήπως μπορούμε να ε, ολοκληρώσουμε κι άλλο ένα σημείο, να δούμε την απαλλαγή μέχρι να έρθει ο Επίτροπος. Ωραία. Ευχαριστώ. Μαζί θα τα πιάσω τα 11 και 12. Καταρχήν να πω ότι η οικονομική πτωτική τάση επηρεάζει και μας και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει λοιπόν να αποδεικνύουμε την καλή διαχείριση των χρημάτων μας ε, και υπέρ της ανάπτυξης ε, η απαλλαγή η λειτουργία της απαλλαγής του Κοινοβουλίου παραμένει ζωτική σε αυτά τα πλαίσια. Στο σχέδιο γνωμοδότησης Αναφέρω την έμφαση στην κατομερισμό εργασίας και στα προβλήματα της βοήθειας. Χρειαζόμαστε καλύτερη, όχι περισσότερη βοήθεια. Θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους οι χορηγοί, να ακούνε τις ε, χώρες εταίρους. Υπήρξε πρόοδος να συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Τώρα ποιος δαπανά τα χρήματα αυτά. Τα, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών είναι οι καλύτεροι, οι πλέον ενδεδειγμένοι ως επιδοπλίστων για να αναλάβουν αυτή τη δουλειά, όχι πάντα όμω. Θα ήθελα η Κομισιόν να σκεφτεί περισσότερο για, για, μια, για κάποιους διάβλους εφαρμογής πιο διαφανείς. Τώρα για τα επισητιστικά θέλουμε καλή ισορροπία μεταξύ διεθνών οργανισμών και άλλων επιλέξιμων ε, φορέων. Το 63-37 ε, κατανομή αυτή μόλις και σέβεται αυτή την ισορροπία. Τώρα για την υγεία και την εκπαίδευση είναι ανήκουστο ε, στον αναπτυγμένο κόσμο να πεθαίνει στη γέννα μια γυναίκα, αλλά στον αναπτυσσόμενο κόσμο πολλές γυναίκες πεθαίνουν κατά τον τοκετό. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μεγαλύτερη προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν. Το AIDS, η ελονοσία, ε, τύφος ε, είναι οδηγούν σε πολλά θύματα και στο παρελθόν και στις διαπραγματεύσεις συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τουλάχιστον το 20% της αναπτυξιακής βοήθειας να το ε, διοχετεύσει στη βασική υγεία και εκπαίδευση. Ο, ε, στήριξη του προϋπολογισμού μπορεί να ε, βοηθήσει ιδιαίτερα σε τομείς όπως η της υγείας και της εκπαίδευσης αλλά όταν είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να δαπανηθούν τα χρήματα εκεί που πρέπει το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε αδυναμίες, σφάλωτα στις πληρωμές. Ε, θα πρέπει να, να επαληθεύεται η τήρηση των όρων. Ε, καλό είναι λοιπόν η Κομισιόν να έχει συστήματα ελέγχου και ε, επιτήρησης και μετά να, δίνει, ε, να παρακολουθεί μέχρι τέλους της, συν, τη συνέχιση της βοήθειας. Επίσης πρέπει να βοηθήσουμε στη δημιουργία ικανοτήτων. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν ε, διότι το ε, υπήρξαν επίπεδα ρεκόρ στο 2008 για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτό ε, υπάρχουν όμως και προβλήματα προσωπικού και κάποιες άλλες τις αδυναμίες που κατεπηγόντως πρέπει να εξετάσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Μάρτιν Τένιγκτον πριν υποδεχθούμε τον Επίτροπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος. Ε, χαιρετίζομαι την έκθεση του εισηγητή. Επιτελέσαμε πρόοδο σε πολλά θέματα που έθεσε το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα εκδίδουμε κατευθυντήριε γραμμές για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ε, ε, διάβλους ε, ώστε οι ΜΚΟ να διαχειρίζονται τα χρήματα, κονδύλια που του στέλνουμε πιο αποτελεσματικά. Επίσης κάνουμε αναθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών μας ελέγχου ε, αυτά τα πράγματα που αναφέρουν στην έκθεσή τους στο ελεγκτικό συνέδριο τα παρακολουθούμε και θέλουμε να ανταποκριθούμε. Ε, βεβαίως προσέχουμε ιδιαίτερα αυτά που αναφέρονται για τον προϋπολογισμό, τη δημοσιονομική στήριξη ε, από το ελεγκτικό συνέδριο Ε, πήραμε ενθαρρυντικά μηνύματα από το ελεκτικό συνέδριο σχετικά με το πώς τεκμηριώνουμε τώρα τις αποφάσεις μας σχετικά με την δημοσιονομική στήριξη και τις πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης. Τώρα, για ε, τους οργανισμούς Ηνωμένων Εθνών κάναμε μια αξιολόγηση πριν από λίγο καιρό και το αποτέλεσμα ήταν ότι δώσαμε οδηγίες πέρσι τον Ιούνιο ε, απογεγραμμένες από τον Λουί Μισελ σχετικά με τους διεθνείς οργανισμούς και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Τα πάντα πρέπει να τεκμηριώνονται, να καταγράφονται και να είναι σαφές γιατί είναι αυτό, γιατί είναι αυτή το πιο κατάλληλο κανάλι ή διάβλος ε, για την ε, παράδοση της βοήθειας. Σε ό,τι αφορά τώρα το, τη στενότητα στο προσωπικό, καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες σας, υπάρχουν κάποια θέματα που πάμε να λύσουμε. Ε, αυτά έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις, ε, τους επισυμβάσει υπαλλήλου. Συνεργαζόμαστε και με άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν για να λύσουμε τα θέματα αυτά. Και τέλος ε, επανέρχομαι στο ζήτημα του 20% Εμεί υποβάλλουμε εκθέσεις σε τακτά διαστήματα πάνω σε αυτό το θέμα και ο κύριο Μισελ νομίζω ότι από την επιστολή πέρσι στην Επιτροπή με πολύ λεπτομερή ε, περιγραφή της κατάστασης και κατανομή μέχρι το 2007 τα στοιχεία για το 2008 και το 2009 είναι πολύ ενθαρρυντικά ε, ο καταμερισμός ήταν 20% ε, στα πλαίσια του DCI ε, και το 2009 θα είναι πολύ υψηλότερο, οπότε ε, βλέπετε τις αυξημένε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Όπως και παλιότερα σας διαβεβαιώνω και αυτή τη φορά ότι είναι υποέλεγχο η κατάσταση, κατανοούμε τις ανησυχίες της Επιτροπής σας και ανταποκρινόμεθα σε αυτές. Αν, αν υπάρχουν από τον εισηγητή και άλλα κάποια θέματα που θέλει να ε, θέσει ακόμη, ε, μπορώ ευχαρίστως να προσπαθήσω να απαντήσω. Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, 5 το απόγευμα, είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ο κύριος Μίτσελ της Κομισιόν, δεν θέλω να καθυστερήσω τώρα, αλλά μας στείλει μια, ε, ένα σημείωμα σχετικά με την ε, χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί πολλοί πολίτες μας ταξιδεύουν εκεί και καλό είναι να βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούν τα προγράμματα αυτά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο Ανάπτυξη, κ. Πίμπαλ, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω την περασμένη εβδομάδα στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Ανάπτυξη στην Ισπανία. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Επιτροπή μας ο κύριος Πίμπαλξ από την ακρόασή του ως Επιτρόπου Αρμόδιου, ω υποψήφιο Επιτρόπου στις 11 Ιανουαρίου. Τον ευχαριστούμε για την τον συγχαίρουμε για την ε, εκλογή του και τον ευχαριστούμε που ήρθε τόσο γρήγορα ενώπιον μας αμέσως μετά την ε, ανάληψη της, των ε, αρμοδιοτήτων του. Ο κ. Πίμπαλξ θα παρουσιάσει τι προτεραιότητε για το, στον τομέα τη ανάπτυξη επόμενους μήνες και θα θέλαμε την ίδια ευκαιρία να εξετάσουμε και κάποιε δεσμεύσει που είχε αναλάβει ο κ. Πίμπαλξ στην ακρόασή του, ιδιαίτερα σε διαφορά τους του στόχου τη τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια. Κύριε Πίμπαλξ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και που με καλέσατε. Και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας ότι μπορώ όντως να διαχειριστώ αυτό το τομέα. Θα είναι πραγματικά ανηφορικός ο δρόμος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Έρχομαι από το Συμβούλιο όπου συζητήσαμε πολλά πολιτικά θέματα για να τηρήσουμε διάφορες δεσμεύσεις, όπως ε, τις έθεσε και ο πρόεδρος. Θα ακολουθήσουν λοιπόν όλες οι, ε, ε, όλες οι πολιτικές. Συζητήσαμε και την ΑΕΤ με τους Υπουργούς Εξωτερικών και επίσης είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος επιτρόπος για την ΕΤΚΟ για όλα τα θέματα που αφορούν και τις θεωρήσεις και όλα αυτά βεβαίως γίνονται σε, από κοινού με τους συναδέλφους μου. Οπότε θα ακολουθήσουμε πραγματικά την ε, γραμμή αυτή που σας υποσχέθηκα όταν ήμουν εδώ. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν τίποτα. Τα θέματα που σχετίζονται με τις εξωτερικές σχέσεις ανισχύονται ε, όλο και περισσότερο θα έχουμε μια ομάδα επιτρόπων ε, να συζητήσει τα θέματα αυτά το Μάρτι και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του ε, Μαρτίου, αν θέλετε, μπορώ να ξαναέρθω στην Επιτροπή σας και να σας αναφέρω ε, ποιες είναι οι προτάσεις έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι ό,τι και να κάνουμε δεν θα διακυβεύσουμε την α, αναπτυξιακή βοήθεια. Βεβαίως, εγώ ευχαρίστω να σας α, τηρώ ενήμερους. Από τις 11 Μαρτίου και μετά θα υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τις ε, απτές προτάσεις, γιατί ως τότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση στην Κορεπέρ. Και η συζήτηση στην Κορεπέρ είναι το τέλος της διαδικασίας, όχι η αρχή. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ ακόμη, γιατί έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Πιστεύω ότι η Ισπανική Προεδρία ε, τα έχει πάει πολύ καλά και βασική, στόχη ήταν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για δύο βασικά θέματα. Και επειδή επιβεβαίωσαν αυτά που περίμενα κι εγώ, ότι δηλαδή πρώτον η αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας είναι η ιερία γελάδα και για το Συμβούλιο, οπότε όλα τα κρατημέλη έχουν δεσμευτεί ότι ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Καμία χώρα δεν ήταν αντίθετη. Δεύτερον, άλλη δέσμευση. Λάβαμε κάποιες πληροφορίες για, από τον ΟΣΑ. Όλες οι χώρες όμως ε, επιβεβαίωσαν ότι θα τιμήσουν τις ε, υποχρεώσεις τους για το 2015, για το 0,7 δηλαδή, για την Ευρώπη των 15 και για 0,3 για την Ευρώπη των 12. Είναι μεγάλη ευθύνη λοιπόν για μένα και την Άνοιξη θα προσπαθήσουμε με ένα συγκεκριμένο πακέτο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και με μία μόνιμη παρακολούθηση του θέματος. Τώρα, αν δεν τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες ε, ε, δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα τα οποία θα μας εγγυούνται την επιτυχία. Γιατί για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανανεώσιμες ειδικά, χάσαμε. Δεν επιτύχαμε έναν από τους στόχους για το 2010. Δεν τον έχουμε επιτύχει. Και επί τη βάση αυτού αυτό ήταν ένα βασικό επιχείρημα που είπαμε ότι πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα αυτοκίνητα. Καταλήξαμε σε δεσμευτική νομοθεσία γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία δεν, κατα, δεν επέτυχε το στόχο τη. Οπότε, αν δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω πως θα πρέπει να σκεφτούμε μια νομική πρωτοβουλία. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να είναι με διαφορετική μορφή. Μπορεί να είναι κοινοτικό φόρο, μπορεί να είναι κοινοτική χρηματοδότηση, μπορεί να είναι εθνική νομοθεσία, δεσμευτική. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δούμε ε, σε περίπτωση που δεν, ε, ε, δεν επιτύχουμε τον στόχο μας και πώς θα κυλήσει το 2011. Τώρα, για το αερινό πακέτο. Για το ειρηνό πακέτο έχουμε δύο ανακοινώσεις, τρεις ανακοινώσεις, μία γενική για το πώς προχωρούμε προς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και για άλλα θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε λοιπόν δύο ανακοινώσεις και έχουμε και δύο έγγραφα εργασία για την εκπαίδευση και για την, ε, για την ισότητα των δύο φύλων. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το γραφείο μου το παρακολουθεί και τα έγγραφα αυτά πιστεύω ότι θα, έχουν πραγματικά, θα είναι πραγματικά ποιοτικά, ώστε και το Συμβούλιο Εξωτερικών να μπορεί να συμμετάσχει το, για το Μάη και τον Ιούνιο. και να έχουμε μια συγκεκριμένη ισχυρή θέση της ε, Ευρώπης ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, ώστε να είμαστε ισχυροί και συνεπείς το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ήταν σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου ε, Υπουργών ήταν παρόν ο Δόκτωρ Σαχ, ο νέος διευθυντής του USAID, ο οποίο μας ενημέρωσε ότι και αυτό θα προσπαθήσει ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή η συνεργασία και ο διαχωρισμός, ο καταμερισμός συγγνώμη, των αρμοδιοτήτων. Επίση, συζητήσαμε και άλλα μικρότερα ίσον σημασία θέματα, τα οποία όμω μπορούν να είναι σημαντικά. Το χρονοδιάγραμμα, καταρχήν, γιατί συνήθω. μπορεί να μην βάζουμε συγκεκριμένη πίεση, να μην ασκούμε συγκεκριμένη πίεση σε θεσμικές ε, ε, διατάξεις. Θα υπάρξει ένα έγγραφο από τη Νέα Υόρκη, το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχει καλός σύνδεσμος και με, τον, με το Κοινοβούλιο, αλλά και με την Επιτροπή τη δική σας. ώστε όσοι είναι, ώστε προετοιμάζονται να έχουν ε, μια καλή βάση και σωστή βιβλιογραφία για να το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφής η συνοχή στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού και αυτό πρέπει να γίνει εγκαίρος για να μην πούμε ότι α, τελικά αργήσαμε. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει ε, συνοχή μεταξύ των συζητήσεων στην ε, Βρυξέλλα, στο Στρασβούργο και, το, και την Νέα Υόρκη. Επίσης, προετοιμαζόμαστε για την Συνόδο Κορυφής με την Αφρική Για την Λιβύη επίσης υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ότι θα γίνει 29 και 30 Νοεμβρίου στην Τρίπολη η Σύνοδος Κορυφής, αλλά τώρα υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις θεωρήσεις. Αρκετά περίπλοκα θέματα, προσπαθούμε να τα διαβελευκάνουμε, αλλά σε αυτή τη φάση δεν διακυβεύεται το κατά πόσο θα γίνει ή όχι η Σύνοδος, γιατί πιστεύουμε ότι θα διαλευκανθεί το θέμα γρήγορα. Αλλά Σίγουρα ξέρουμε ότι πρέπει να αντιληφθεί έγκαιρα το θέμα αυτό, γιατί αλλιώ πρέπει να δούμε τι εναλλακτική έχουμε. Οπότε δουλεύουμε και ως προς αυτό. Και τέλος, για την IT, έγινε μια συζήτηση σήμερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και με τον είπα εκπρόσωπο με την ε, συνάδελφο Γεωργίευα έχουμε πολύ καλή ε, συνεργασία, οπότε για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια η βασική πρόκληση είναι το θέμα της στέγασης και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών. Πολλοί συναδελφοί μου έχουν πάει στην ΑΕΤ και στο Πόρτο prince και πέρα από την ε, πρωτεύουσα. Και επίση έχει ξεκινήσει συντονισμό από τα κρατημέλη και την Κομισιόν για αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Σήμερα θα έρθω σε επαφή με δύο πρεσβευτές που ε, αποστέλλονται στην ΑΕΤ για να βοηθήσουν την, το συντονισμό. Και όλοι συμφωνούν ότι η ΑΕΤ είναι πραγματικά ένας, είναι το καλύτερο παράδειγμα για καταμερισμό αρμοδιοτήτων και για συντονισμό. Ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα, προς το παρόν δεν έχουμε όσα αποτελέσματα θα θέλαμε. Η IT λοιπόν είναι πραγματικά μια προτεραιότητα για, την, ε, για μένα και έχω πάρα πολύ καλή υποστήριξη και από τους συναδέλφους και από τις υπηρεσίες της Κομισιόν, ώστε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιφέρουμε πρόοδο. Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Πρέπει καταρχήν να κάνουμε καλή αρχή για, την, για, τους, αξιό, για τους ε, στόχους της, ε, της Πρώτο αυτό και μετά πρέπει να λύσουμε το θέμα της ε, IT. Σαφώς, με σαφή αποτελέσματα και με συνέπεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση εδώ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Χαιρετίζω αυτά που είπε για τους αναπτυξιακού στόχους της χιλιετίας και θα κάνω σύντομα κάποιες παρατηρήσεις κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσω. Καταρχήν θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχής όπως νομίζω έκανα και κατά την ακρόασή σας για το αξίωμά σας ότι η ορατότητα και ο ηγετικό ρόλος στην ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά. Ε, ο Μπόνο, ο Μπομπ Γκέλντοφ, ε, άλλοι συμπατριώτες μου έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν βέβαια, αλλά και η πολιτική επίσης και κάποιος πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο. Θα έλεγα να μιλήσετε με τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή πολιτική της Ένωσης, ούτως ώστε από κοινού να έχετε ένα πρόγραμμα για να μάθει ο Ευρωπαίος πολίτης τι ακριβώς κάνουμε και να δώσει την υποστήριξή του, γιατί είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δέσμευση στην τήρηση και επίτευξη των στόχων και όλα αυτά είναι ορατά. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Επίσης, πολύ σύντομα, σε σχέση με τις εξωτερικές δράσεις, για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων καταρχήν, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό η υπηρεσία αυτή να είναι προσβάσιμη στους ε, ευρωβουλευτές όταν θέλουμε πληροφορίες ή ε, επισκεπτόμεθα της χώρας, της, ε, χώρας. Αυτή η εξωτερική υπηρεσία της Ένωσης θα είναι η εκπροσώπηση. Αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να συνδράμει τους ευρωβουλευτές ε, σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες που επισκεπτόμεθα ή εξετάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό τα μέλη του Κοινοβουλίου να έχουν τη στήριξη που χρειάζονται. Εις ό,τι αφορά τις εξωτερικές δράσεις καθ' αυτές, δεν νομίζω ότι το έγιναν διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ε, οι πληροφορίες είναι από δεύτερο χέρι και θα ήθελα να δούμε περισσότερο τη δανική, δανέζικη πρόταση για τον, ε, οριζόντια, τον οριζόντιο διαχωρισμό. Τώρα οι περισσότερες χώρες είναι υπέρ. Η ε, Πορτογαλία ε, έχει κάποιους δισταγμούς ίσως λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρος είναι Πορτογάλος. Επίσης, για την IT, χαίρομαι με αυτά που είπατε για τον καταμερισμό εργασίας και το συντονισμό. Ε, τώρα που πάμε στην εποχή των βροχών, θα πρέπει να μας διαβεβαιώσετε ότι υπάρχει ένα πλάνο που θα μπορέσει να προλάβει ε, τις ανάγκες. Δεν θα πρέπει μόνο να αντιδρούμε, αλλά να προλαμβάνουμε τις ανάγκες ε, στα πλαίσια της, ε, του καταμερισμού και του συντονισμού. Επίσης, σκεφτείτε, δεν, αναγε, δεν περιμένω να μου απαντήσετε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο ε, ε, ε, αποφάσισε για το 0,7. Άλλοι ξεπέρασαν το 0,7 πιστώσεις υποχρεώσεων. Δεν είναι ρόλο σας να πείτε στα εθνικά κοινοβούλια τι θα κάνουν, αλλά θα μπορείτε να ενθαρρύνετε τις κυβερνήσεις να νομοθετούν, ούτως ώστε όταν αυξάνεται το ΑΕΠ να αυξάνεται η συμβολή και αντίστροφα όταν πέφτει να πέφτει. Όχι όμως να ε, μειώνεται το ΑΕΠ, να μειώνεται η συμβολή και μετά να φέρουν κι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νομοθέτημα σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τις προθεσμίες που θέσατε εσείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ να καλωσορίσω τον ε, νέο Επίτροπο. Ξέρετε κύριε Επίτροπε ότι εμείς στο Κοινοβούλιο εμπιστευόμεθα πάρα πολύ και το πρόσωπό σας και πολλοί από εμάς είπαν ότι εσείς πραγματικά είστε εκείνος που θα επιτελέσει το έργο που πρέπει. Κάποιες ανησυχίες υπάρχουν. Όχι επειδή εσείς κάνατε κάτι αρνητικό, αλλά βλέποντας τη στάση των κυβερνήσεων και της Κομισιόν. Πριν τα πω αυτά, θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω τις προτεραιότητες που μας ε, παραθέσατε και να πω ότι συμφωνώ καταρχήν με τις προτεραιότητες ε, ε, τους στόχους της χιλιετίας, την ΑΕΤ και τις ανακοινώσεις που βεβαίως θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα κάνω πιο πολλά σχόλια. Δεν θα πω επί του παρόντος τίποτε περισσότερο εδώ. Θα περιμένω. Τώρα για τη διακυβέρνηση, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε θέματα αρχής. Εσείς είστε ο αρμόδιος επίτροπος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και επίτροπος υπεύθυνο για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει ελευθερία και επιλογή σε αυτά τα θέματα. Αν μιλήσουμε για αυτές τις βασικές αρχές και αν εσείς ε, ε υπερασπίζεστε αυτές τις αρχές, ε, θα έχετε την απόλυτη υποστήριξη της Επιτροπής μας. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους. Όχι μόνο δηλαδή να δημιουργούν ε, μέσα, εργαλεία που όμως μειώνουν την ορατότητα, που είναι σημαντικό να υπάρχει ε, για να γίνει δεκτή η συνεργασία και η ανάπτυξη, η αναπτυξιακή συνεργασία από την κοινή γνώμη. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε ή να υπονομεύσουμε ε, τη συνεργασία μας. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα μέσα ώστε να ισχύει η αρχή της καταπολέμησης της ε, φτώχειας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα ε, μέσα από τεκμηρίωση ε, συγκεκριμένη. Ε, αν είχαμε 50 κράτη-μέλη, θα καταλάβαινα ότι θα έπρεπε να γίνει επιμερισμός χαρτοφυλακίων, ούτω ώστε να μοιραστεί στα κράτη-μέλη. Αλλά είμαστε 27. 27 κράτη-μέλη και θέλουμε αποτελεσματική πολιτική που πρέπει να είναι και συνεκτική σύμφωνα με τις συνθήκες και εσείς και κανείς άλλος είστε υπεύθυνος για να τα κάνετε όλα αυτά στην πράξη. Πρέπει λοιπόν να ε, ορίσουμε το, την αρχή της καταπολέμησης της ε, στόχες. Μην τα αφήσουμε μόνο στη ρέλεξη. Με κάθε σεβασμό χρειάζεται κάποιος υπεύθυνο για εξωτερικά θέματα, αλλά δεν θα πρέπει να ε, αναφτεθεί το δικό σας καθήκον και έργο σε εξωτερικό φορέα. Ξέρω, εκπήρας, ξέρω τι συμβαίνει τώρα, ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά υπάρχει μια γενικότερη τάση που θέλει να αποδυναμώσει την λειτουργία του επιτρόπου που είναι του αρμόδιου επιτρόπου εν γέννη. Πριν από κάποια χρόνια, κάποιοι από εμά χρειάστηκε να αγωνιστούν για να διατηρηθεί το Συμβούλιο Υπουργών ανάπτυξη. Ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου ήθελε να το καταργήσει. Ε, είχαν ε, πει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε άτυπα συμβούλια Υπουργών Ανάπτυξης, λίγο και συγγνώμη για την έκφραση, σαν να, προσπαθεί, να, να, να προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από μια, κάνοντας πεζοδρόμιο για να μην μπορέσεις να είσαι στο σπίτι σου. Αυτή η προσέγγιση σταμάτησε, αλλά έπαυσε, αλλά συνεχίζεται παρά τα αυτά να εμφανίζεται αν, ε, ανά καιρό. Γιατί να υπάρχει ένας επίτροπος ανάπτυξης όταν ε, όταν έχεις έναν άλλον επίτροπο που είναι αρμόδιος μόνο για την εξωτερική βοήθεια. Στην Επιτροπή, όταν είδαμε τα καινούργια ονόματα της Επιτροπής, ε, είδαμε πολλές, είχαμε πολύ, πολλές περιπτώσεις απογοήτευσης. Συχνά είχαμε την εντύπωση ότι χρειαζόταν εμείς να αγωνιστούμε για να υποστήριξουμε τη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης και δεν θέλω πραγματικά να ε, επιμείνω επιμακρών στο θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για να αναπτύξουμε το χαρτοφυλάκιο της ανάπτυξης στο ιστορικό της Επιτροπής, να δημιουργήσουμε μια ε, πολιτική ανάπτυξης ε, επέκτασης που πρέπει να έχει πλήρη συνέπεια στις συναντήσεις του συντονισμού. Ξέρετε ότι θα έχετε δύσκολη δουλειά γιατί θα χρειαστεί να αναπτύξετε ε, μια σειρά θεωρητικών ε, θέσεων στο εσωτερικό της Επιτροπής. Εάν θέλετε λοιπόν την υποστήριξη πρέπει να συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ε, φτωχών και των άμυρων του κόσμου. Εάν αγωνιστείτε για τις θέσεις σας, θα έχετε την επιτροπή μας μαζί σας. Το λέω αυτό χωρίς να έχω συζητήσει με τους συναδέλφους, αλλά είμαι σίγουρος ότι ένας βασικός πόλος της εξωτερικής δράσης της Ένωσης ήταν η πολιτική ανάπτυξη, ιδίω για τις, χώρες, για χώρες και εν πολλής χάρη στην καλή συνεργασία Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα Επιτροπή Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου και, ε, το και του, του χαρτοφυλακίου που έχετε εσείς. Ευχαριστώ. Thank you. Κυρία Κέλλερ, έχω πολλές ερωτήσεις. Τρεις θα κάνω όμως μόνο. Θα μιλήσω για ένα θέμα που συζητήσαμε προηγουμένω. Η συνεκτικότητα των πολιτικών στον τομέα τη ανάπτυξη. Είπατε ότι είναι μία από τι προτεραιότητε που θέλετε να θέσετε. Περισσότερο συμφωνούμε. Έχετε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα βελτιώσει την κατάσταση έχετε εξετάσει, θα εξετάσετε στο μέλλον τις προτάσεις που υποβάλλουμε στο σχέδιο έκθεσης. Δεν ψηφίστηκε εμένα, αλλά υπάρχουν προτάσεις προς την Επιτροπή. Επίσης, εξετάσετε ή θα εξετάσετε στο μέλλον την πρόταση που κάναμε για το μηχανισμό καταγγελιών, όταν είχαμε προτείνει ο διαμεσολαβητής να εξετάζει καταγγελίες για ασυνέπεια πολιτικών. Δεύτερο, Αυτά που είπε και ο κύριος Γκέρενς, προγραμματισμός και εφαρμογή, και των αναπτυξιακών, της αναπτυξιακής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Πολλά από αυτά δεν έχουν μπει στο δικό σας χαρτοφυλάκι. Μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είπατε ότι θα, τρίτο, θα προσπαθήσετε να τηρήσουν τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη το ποσοστό του 0,7%. Τι θα κάνετε ακριβώς για την επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την αλλαγή του κλίματος, την προσαρμογή των χωρών και το μετριασμό των συνεπειών του κλίματος. Γιατί κάποια κράτη, π.χ. η Γερμανία, είχε πει ότι θα βγάλει το κονδύλι αυτό από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Τι λέτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίμπαλξ για να απαντήσει σε αυτές τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Well, thank you very much. Ευχαριστώ. Yeah, sorry, sorry. For visibility on leadership, I Τώρα, πόσο ορατοί θα είμαστε. Συμφωνώ ότι μόνο με μεγαλύτερη ορατότητα θα μειωθεί η φθήνουσα πορεία της αναπτυξιακής πολιτικής. Μίλησα τώρα σήμερα με δημοσιογράφους ε, ε, από τις νέες χώρες και όταν μιλάμε για φτώχεια, ε, συνήθως με ρωτάνε γιατί τη φτώχεια, νομίζουν ότι ασχολούμαι με θέματα ανάπτυξης στο εσωτερικό των κρατών φτωχούς δηλαδή μέσα στα κράτη-μέλη. Τους λέω δεν είναι αυτό το πράγμα. Ε, χρειάζεται να το κάνω για να μπορέσω να ενισχύσω την επικοινωνία στο εσωτερικό της Ένωσης ιδιαίτερα. Στο εσωτερικό της Ένωσης έχουμε γραφεία της Επιτροπής έχουμε προπολογισμό. Θα ζητήσω από τη συνάδελφο κύριε Ρέντινγκ να με βοηθήσει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Οι αντιπροσωπείες εξωτερικής δράσης, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι δεν πάμε πίσω, μόνο μπροστά θα πάμε. Και αυτή τη στιγμή υπήρξε ε, συνεργασία μεταξύ αντιπροσωπιών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Μπορεί να μην ήταν πάντα τέλειες οι σχέσεις, αλλά γενικά είχαν επιτυχή ιστορικό, επιτυχές ιστορικό. Ε, εκεί που υπήρχε επίσκεψη του Κοινοβουλίου, ας πούμε, το αναλάμβανε η Επιτροπή και το, και το προχωρούσε και με, ε, επιτυχή, με το, το πετύχαινε καλά. Τώρα για το splitting στο Συμβούλιο. Εγώ διαβάζω προσεκτικά τη συνθήκη και λέει Καταρχάς, προτάσει της είπα της εκπροσώπου. Αυτή υποβάλλει την πρόταση. Κατόπιν συμφωνεί Επιτροπή. Και εγώ δηλαδή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ε, κατά πλειοψηφία, αλλά γενικά η συμφωνία απαιτεί συνένεση. Κατόπιν είναι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο μια τυπική διαδικασία. Και κατόπιν ομοφωνία στο Συμβούλιο. Κάτι που σημαίνει ότι και υπό το Γαλλία, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι από εκεί, θα μπορεί να επηρεάσει πολύ. Και ούτω ή άλλω αυτό ξεκινάει με μια άτυπη βολιδοσκόπηση στο εσωτερικό τη Κορεπέρα. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριο Γκέρεντ μας ρωτήθηκε, με ρωτήθηκα κατά τη διάρκεια της ακρόαση. πού είναι η γραμμή, πού λες ότι χάσαμε. Όντως υπάρχει κάποια ε, φάση, κάποιο χρονικό, κάποια, στιγμή που ε, μπορεί να πεις ότι η πολιτική αποδυναμώθηκε, αλλά εγώ νομίζω ότι στο εσωτερικό της Επιτροπής ε, υπάρχει μια πλήρης βούληση αύξησης και, αν, και ενίσχυσης και όχι αποδυνάμωσης της πολιτικής ε, ε, της πολιτικής για την ανάπτυξη. Και η συνθήκη λέει ότι μόνο ο ύπατος εκπρόσωπος εκπροσωπεί τη σχέση, την επιτροπή στη σχέση της με τις τρίτες χώρες. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι θα μπορούσα να ξεχάσω τη χαρά του να έχω πολιτική συζήτηση εγώ προσωπικά. Δεν λέει η συνθήκη όμως ότι θα πρέπει να αποδυναμωθεί η συγκεκριμένη πολιτική, που σημαίνει ότι η πολιτική, ε, ο πολιτικός διάλογος υπό την αιγίδα της υπό της εκπροσώπου σημαίνει ότι η πολιτική ανάπτυξη θα αποδυναμωθεί. Δεν θα... Τώρα, για τι ερωτήσει που θέσετε για τα κράτη-μέλη, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχολιασμό για την άποψη που έχει το Α ή το Β κράτο μέλο. Η συζήτηση είναι μπροστά μα, δεν είναι πίσω μα για την ανάγκη να έχουμε μια διενεργή προσέγγιση στην ε, στέγαση. ναι, έχουμε. Έχουμε όλες τις δυνατότητες και έχουμε και τη δυνατότητα για τη δημιουργία καταφυγίων ε, στην ε, IT. Σε ό,τι αφορά την Ένωση λοιπόν, δεν θεωρώ ότι έχει αποδυναμωθεί η προσέγγιση μας στην παροχή στέγης. Βεβαίως η κυρία είναι η αρμόδια η οποία θα μπορεί να απαντήσει, η οποία μπορεί να απαντήσει τι πήγε. Είμαστε σε θέση να χτίσουμε στέγη για 100.000 ανθρώπους. Δεν μπορώ να σας το πω, αλλά μόλις γυρίσει θα σας απαντήσει. Πάντως έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Έχουμε συγκεκριμένη έμφαση στην ανθρωπιστική ενέργεια, ε, στην ανθρωπιστική προσέγγιση. Τώρα για τη Βρετανική νομοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι νόμο ε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ε, νομίζω ότι μόνο νομοθετικά ε, μπορεί να το επιλύσουμε με, με, με, κοινοβουλευτική κυριαρχία και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπο και ο ευκολότερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το πρίτημα. Αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, επικριτικές φωνές. Δεν ξέρω βέβαια αν πέρασε αυτό στο κοινοβούλιο τη μεγάλη Βρετανία. Υποβλήθηκε το σχέδιο αλλά δεν έχω λάβει ακόμα επιβεβαίωση ότι εγκρίθηκε. Για τα σχόλια Γκέρενς, για τα θέματα διακυβέρνηση του ιστορικού τη ε, επιτροπή, απάντησα εν μέρη. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω που πιστεύω ότι ενισχύουν τις θέσεις μου, δεν τις ε, αποδυναμώνουν. Και εγώ και η κυρία Τέλο η παρουσία τη κυρία Γεωργίου δεν με αποδυναμώνει, με ενισχύει πιστεύω, διότι ε, ε, μαζί δουλεύουμε, με υποστηρίζει και πιστεύω ότι η ΕΚΟ, η ΕΚΟ είναι μία δομή που μπορεί να που αισθανόταν ότι ήταν παραμελημένη και τώρα αισθάνεται ότι την, ε, τη βλέπουν, την παρακολουθούν, θέλουν να καταλάβουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι, όλα, ότι αυτή η αλλαγή μας ενισχύει, δεν μας αποδυναμώνει. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κρίμα πως, ε, που δεν υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών ανάπτυξη, όντω το άτυπο είναι ε, βραβείο Αλλά και άλλα συμβούλια καταργήθηκαν πιο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε το ρόλο των πολιτικών ανάπτυξη, και εδώ θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ε, λέτε ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο την Επιτροπή. Ε, στο εσωτερικό της Επιτροπής. Κοίταξτε, δεν είμαστε και πολύ καινούργοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο κάνουμε μια συζήτηση για την Ευρώπη του 2020. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε αρκετά πράγματα. Ε, και νομίζω ότι είναι κατανοητό εν γέννη ότι δεν μπορείς να έχεις συνοχή στην πολιτική αν δεν έχεις μια προσέγγιση παρόμοια σε όλους τους τομείς. δεν μπορεί να είναι μόνο δηλαδή οικονομική η προσέγγιση μας. Ξέρω το μηχανισμό καταγγελιών που προτείνεται. Θα μελετήσω την ε, έκθεσή σας. Δεν θέλω να λάβω θέση προς το παρόν. Αξίζει να το συζητήσουμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Αλλά μία έκθεση, ακόμα και, σε... και σχέδιο έκθεση, είναι θετικό γιατί καταλαβαίνω τι θέλετε να συζητήσουμε και τι προτάσεις να υποβάλουμε. Για το... την αναπτυξιακή βοήθεια και το EDF είναι σαφές ότι κατά την ε, ε, δική μου θητεία η ένταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προπολογισμό δεν είναι εφικτή. Ε, βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρουμε πιο κοντά τις αρχές του προγραμματισμού. Όσο πιο κοντά δέχεται τα θέματα αυτά στη διαφάνεια γίνεται. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, να συνεχίσουμε δηλαδή να ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση αλλά μια απόλυτα ενιαία προσέγγιση δεν είναι δυνατή. Τουλάχιστον τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη περίοδο όταν θα υπάρξει πραγματική ένταξη του EDF στον ε, προπολογισμό. Αλλαγή κλίματο. Δεν άλλαξε η θέση μου. Η βοήθεια, η υπόσχεση βοήθεια δόθηκε, δόθηκε πριν την αλλαγή του κλίματο, οπότε ό,τι δώσουμε για το κλίμα είναι εξτρά. Μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει τα κράτη-μέλη Πιστεύω ότι στην αλλαγή του κλίματος, η αλλαγή του κλίματος είναι μια συζήτηση που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στο Μεξικό, πρέπει να μην ανακατεύουμε τα δύο θέματα. Γιατί αν τα ανακατέψουμε θα αποτύχουμε και στην ανάπτυξη και στην Νέα Υόρκη και στο Μεξικό. Αυτό σημαίνει ότι για του πολιτικού μα στόχου δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια, γιατί κανεί δεν το πιστεύει. Οι εταίροι μα ιδίω. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπαγρυπνούμε, αλλά σήμερα δεν έχω καμία ένδειξη ότι γίνεται προσπάθεια από κάποια κράτη να, καταστρατηγήσει τις, ε, να καταστρατηγήσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν γίνεται ακόμα παιχνίδι με τα νούμερα, τουλάχιστον όχι στη φάση αυτή. We have three more speakers. Τρεις ομιλητές ακόμη έχουμε. Η κυρία Σνίμπαρ Γιάστραμ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Θυμάμαι πολύ καλά την καλή σας και καλά προετοιμασμένη παρουσία σας εδώ, την εμφάνισή σας και θυμάμαι και ορισμένα από αυτά που μας είπατε τότε. Κατά την ακρόασή σας αναφέρατε ότι το θέμα του αντίκτυπου των επενδύσεων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων μη ευρωπαϊκών δρόντων, κυρίως Κίνα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Αφρική, θέλατε να το ε, θεωρήσετε προτεραιότητα. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι μη Ευρωπαίοι ε, παρεμβαίνοντες επενδυτές, Κινέζοι κυρίως στην Αφρική, σε ποιο βαθμό μπορούν να συνεργαστούν στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε ποιο βαθμό θα υπάρξει συμφωνία για τους στόχους, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάζεται για κάποιον ανταγωνισμό για αυτούς τους ε, νέους επενδυτές και πώς κρίνεται το γεγονός ότι σήμερα Κινέζοι όπως και ε, Άραβες ε, επενδυτές και άλλα ιδιωτικά ε, funds πολλές φορές κάτω από αμφίβολες συνθήκες αγοράζουν μεγάλες, ποσότη, μεγάλες εκτάσεις γεών ούτως ώστε να προχωρήσουν μετά ε, σε εξαγωγές ή να αντισταθμίσουν ε, εξαγωγές ε, με την αγορά αυτήν. Πολλές φορές δηλαδή ορισμένοι εξάγουν τις, τα τρόφιμα, άλλοι κάνουν την προσπάθεια να τις διοχετεύσουν προς τις δικές τους χώρες. Ο κύριος ευχαριστώ. Δεν είχα τη δυνατότητα και Επίτροπε να ήμουν παρόν στην ακροασή σας γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε μία από τις πέντε ημέρες χιονοπτώσεων της Μαδρίτης φέτος που δείχνει ότι η αλλαγή του κλίματος είναι εμφανέστατο πλέον φαινόμενο. Θα ήθελα να μιλήσω για τρία θέματα. Το ένα είναι η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Το δεύτερο, οι στόχοι της χιλιετίας. Και το τρίτο, θέλω να επανέλθω στην θεσμική διάθεση. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, νομίζω ότι κομμάτι της δουλειά σας είναι να μην να αποφύγετε τον καταγγελματισμό, να συντονίσετε καλύτερα τους δωρητές και να επιτύχετε μια καλύτερη κατανομή εργασίας μεταξύ της Ένωσης, των υπηρεσιών της Ένωσης και των κρατών μελών γίνεται όλο ένα και περισσότερο σαφέ ότι η αποτελεσματικότητα τη βοήθεια και ο τρόπο που τη διαχειριζόμαστε είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για να πετύχουμε του στόχου που με τη βοήθεια αυτή θέλουμε να πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά του στόχου τη χιλιετία, η εντολή σα και η δική μα λύγει το 2014. Το 2014 είναι τα σύνορα της περίοδου κατά την οποία πρέπει να τηρήσουμε τους στόχους που θέσαμε το 2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το 60% της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο, έχει μία υποχρέωση, μία ευθύνη, ένα καθήκον, να επιτύχει μέχρι το 2015 οι χώρες της Ένωσης να τηρήσουν τους, τις δεσμεύσεις τους και πριν το 2015 να θέσουμε ένα νέο ορίζοντα, ένα νέο σύνορο, νέες δεσμεύσεις και την υποχρέωση να, όπως είπα, ορίσουμε ποιο είναι αυτό το νέο σύνορο, σύνορο ποιες είναι οι νέες δεσμεύσεις μετά το 2015. Ζητώ λοιπόν να είσαστε ενεργός στον καθορισμό των στόχων αυτών, όπου σίγουρα το Κοινοβούλιο, Επιτροπή και η Επιτροπή θα σχηματίσουν μια στρατηγική συμμαχία για να παρατείνουν τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θεσμική διάρθρωση, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο που δεν το έχετε ακούσει συχνά. Συνήθως θα σας λένε να υπερασπίζεστε με νύχια και με δόντια μέχρι θανάτου τις αρμοδιότητες στο εσωτερικό της Επιτροπής. Να αντιστέκεστε σε άλλους φορείς της Επιτροπής που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, να υποστηρίζετε την αυτονομία σας, να εμποδίζετε. Εγώ σας ζητώ κάτι διαφορετικό, όχι το ανάποδο. Όχι μόνο να υπερασπιστείτε την αυτονομία σας, αλλά να προσπαθήσετε να περάσετε στην υπόλοιπη επιτροπή της θέσης σας. Το φρούριο του Επιτρόπου Ανάπτυξης είναι περισσότερο στέρεο αν μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την Επιτροπή, όλες τις γενικές αποφάσεις της Επιτροπής, τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και το ρόλο του Κοινοβουλίου, παρά αν εσείς αγωνίζεστε με πάθος να υπερασπιστείτε το δικό σας κομματάκι των αρμοδιοτήτων. Εγώ, λοιπόν, θα σας ζητώ να περάσετε, να σπρώξετε, να ρίξετε σαν χιόνι πάνω από, την, ε, ε, από τις υπόλοιπες των επιτροπών το θέμα της ανάπτυξης. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα αυτό συζητήθηκε εν μέρη. Αλλά επειδή όταν ήμουν, είχα πάει στην Αγκόλα το Δεκέμβριο ε, για τις εργασίες ΑΚΕ και επισκέφτηκα μια σειρά περιοχών και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από κάποιες περιοχές που μου είχαν πει ότι ήταν τα πιο ενεργά κέντρα ανοικοδόμηση και ανάπτυξης τη χώρα. Στην περιοχή αυτή, στις περιοχέ αυτέ, που ήταν τεράστια εργοτάξια, δρόμοι, κέντρα, διαπίστωσα με εντύπωση ότι το εργατικό δυναμικό που δουλεύει ήταν εκατοντάδες αποκλειστικά όμως Κινέζοι κάθε επίπεδο ε, από το μπετατζή μέχρι το μηχανικό Μόνο Κινέζοι. Δούλευαν στα εργοτάξια, είχαν φτιάξει δικά τους κέντρα εγκατάσταση. Εγώ διαπίστωσα ότι ο πληθυσμό ζει στο δρόμο, Υπάρχει μια περιοχή που, είναι πραγματικά μια χωματερή που μένει ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να βοηθήσει το πληθυσμό των αφρικανικών χωρών στα αναπτυξιακά έργα που προσπαθούν να εφαρμόσουν. Μπορεί να κάνει κάτι η Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Well, uh, Mrs. Περίπου οι δύο κυρίες τα ίδια ερωτήματα έθεσαν. Το θέμα είναι όμως κυρίως ποιε είναι οι σχέσεις με τον εαυτό μα κυρίως και μετά οι σχέσεις μας με τους Κινέζους. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ισχυρή και ενωμένη στην, στα θέματα αναπτυξιακή βοήθειας. Ε, συντονισμός λοιπόν, μερισμός εργασία είναι βασικά. Πρέπει λοιπόν να μην θεωρούμαστε 16 δωρητέ, 15, 28, αλλά ένα δωρητή με όλες αυτές τις υπηρεσίες που συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Καταρχήν πρέπει να είμαστε ισχυροί και ορατοί, να φαίνεται το τι κάνουμε. Να θεωρούμε θα ένας Ευρωπαίος δωρητής. Και η IT μα δίνει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πράξουμε αυτό και πρέπει να την ε, χρησιμοποιήσουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι ακόμη πρέπει να συζητήσουμε και με το Κοινοβούλιο αλλά και με την κοινωνία για το πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Βέβαια, εντάξει, ω ε, επίτροπο θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικό στο πώ χρησιμοποιώ τι λέξει. Αλλά το θέμα είναι πώ θα διαχειριστούμε το θέμα αυτό τη αντίθεση μεταξύ των υποδομών του, του προπολογισμού, τη δημιουργία ε, δυναμικού, δυνατοτήτων. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά και δρούμε και σε, ό, και σε όλους αυτούς τους τομείς. Δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε ή το ένα ή το άλλο. Κάνουμε πολλά λοιπόν ταυτόχρονα και ίσως έτσι αποδυναμώνουμε και τους εαυτούς μας. Οπότε σε ένα βάθος χρόνου θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ας πούμε την, ε, την ε, ένδυα. Αν το κάνουμε αυτό, θεωρώ ότι θα είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να δούμε και το θέμα της ε, Κίνας. Οι Κινέζοι, το να βοηθούν οι Κινέζοι τον αναπτυσσόμενο κόσμο, εντάξει, είναι θετικό. Αλλά αν τελικά το, τα ωφέλη είναι λιγότερα από τα προβλήματα, τότε θα πρέπει να το δούμε. Εμεί θα πρέπει πάντως να μείνουμε παρα... ε, σταθεροί στι αρχές μας. Αν κάποιος έχει αντίθετα ε, επιχειρήματα, εντάξει μπορεί να έρθει και να μας πει όχι εσείς δεν κάνετε καλή δουλειά, αλλά τουλάχιστον εμείς πρέπει να έχουμε σαφή ε, στοχοθέτηση. Πρέπει να δείξουμε ποια είναι η δική μας διάθεση, ότι δηλαδή οι δικές μας πολιτικές είναι ισχυρές που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αξιοπιστία κτλ. Για το θέμα των ε, θέσεων εργασία είναι σημαντικό. Δεν είναι θέμα ε, τη αναπτυξιακή πολιτική να δώσει δουλειά στην ε, Αφρική ή σε άλλε αναπτυσσόμενε χώρε. Το βασικό θέμα τη πολιτική και από κοινού με τον ε, ΟΗΕ και με τους Κινέζους, για την ΑΕΤ τουλάχιστον, είναι να δώσουμε τους, ε, τις θέσεις εργασίας στους ΑΕΤΙΝΟΥΣ. Να τους δώσουμε δηλαδή την αίσθηση ότι έχουν αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι σημαντικό να το ακολουθήσουμε. Εγώ θα είμαι ανοιχτό με τους Κινέζους και θα τους πω ότι εγώ πιστεύω ως Επίτροπος ε, Ανάπτυξη ότι δεν ε, δίνεται αρκετή, ότι δεν αξίζει τον κόπο. Ακόμη βέβαια διαβάζω την ε, πολύ καλή έκθεση της ε, Υπηρεσίας Ανάπτυξης στο, της Νορβηγίας για τους φορολογικούς παραδείσους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο από, αυτή την, από την έκθεση του 2001 που λέει ότι η καλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη είναι να επενδύσουμε στην δημιουργία δυνατοτήτων. Γιατί έτσι αξίζει τον κόπο να υπάρχουν αυτέ οι υποδομέ. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε αυτό και νομίζω ότι και η Κοκομπού θα πρέπει να μα βοηθήσει και να πούμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Ξέρουμε ποια είναι τα ρίσκα, αλλά θα προχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από τα πράγματα που οι Κινέζοι θεωρούμε ότι κάνουν καλύτερα και παρόλα αυτά να μπορούμε να τους επικρίνουμε όταν θεωρούμε ότι η πολιτική τους δεν είναι ενδεδειγμένη. Δεν χρειάζεται να αντεπόμαστε επειδή κατακρίνουμε τους ε, ε, Κινέζους για τα θέματα που έθιξε ο κύριος Γκερέρο. Ακόμα είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Η Ισπανική Προεδρία και η Επιτροπή προετοιμάζει τους καταλόγους, τους πίνακες με τους ε, σημαντικούς ή λιγότερο σημαντικούς ε, δωρητές. Αλλά ε, έχουμε κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ καλές, με πολύ σωστή δηλαδή κατανομή αρμοδιοτήτων και κάποιες άλλες περιπτώσεις για, την, για τις οποίες δεν δίνουμε την απαραίτητη βοήθεια. Οπότε αν εξελίξουμε αυτή τη στρατηγική, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Οπότε στα χέρια μας είναι, στις πολιτική, στην πολιτική μας επαφή, να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για το μετά το 2015. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Γιατί αν αρχίσει κανείς την συζήτηση για το μετά το 2015, το, κίν, το κίνδυνο είναι ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι στόχοι μέχρι το 2015 και η συζήτηση για, αυτό το, για αυτή την χρονική περίοδο θα πρέπει να γίνει. Αλλά όχι αντιγράφοντας τους αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας, είναι σημαντικό να, έχουμε, να θέσουμε συγκεκριμένε δεσμεύσεις, συγκεκριμένου συντονισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά να μην προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε του ε, στόχου τη χιλιετία και να πούμε ότι να, μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουμε του ίδιου στόχου, απλώ με λίγο υψηλότερα ποσοστά. Πρέπει να κάνουμε δι, μια καινούργια συζήτηση. Νέα, διαφορετική ποιότητα συζήτηση. Να μην ε, μπλέκουμε τα δύο πράγματα. Ο κόσμο του ή άλλω δεν σταματάει το 2015. Τώρα και τα θεσμικά. Ε, εγώ, ο, θεσμικό μου, ο θεσμικός μου ρόλος είναι αρκετά ισόρροπος. Εγώ είμαι στο, ήμουν στο πρώτο συμβούλιο, οπότε σε οποιαδήποτε συζήτηση θα πρέπει να είμαι σε θέση να θέτω πάντα το θέμα την πτυχή της ανάπτυξης. Συμμετάχοντας λοιπόν σε αυτό το συμβούλιο, δεν υπήρξε άλλο συμβούλιο για την ανάπτυξη, οπότε ήταν η κατάλληλη θέση μου να είμαι εκεί. Και επίσης, σε συνεργασία με την κυρία Άστον, πάντα βάζουμε στην ατζέντα θέματα ανάπτυξης. Επίσης, το θέμα τώρα είναι η, που πάσχει είναι η διαδικασία ολόκληρη. Πώς δηλαδή μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να ρυθμίζουμε τις λεπτομέρειες με τις αντιπροσωπείες. Και επίσης έχω την πλήρη ευθύνη της ΕΤΚΟ, που ποτέ δεν υπήρχε παλαιότερα. Και αυτό καλύπτει και τις ε, χώρες του ε, μηχανισμού και του ταμείου, αλλά και της νέας ε, πολιτικής γειτονίας. Είναι λοιπόν μια πλήρης διαδικασία. Οπότε, σε ένα βαθμό, έχω μια καλή γενική εικόνα το που πάν, του που πάνε τα χρήματα, ή τέλος πάντων η υπηρεσία μου έχει, και αυτό νομίζω ότι ενισχύει την όλη διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ε, συνενώσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία και χρειαζόμαστε βέβαια και την δική μας, τη δική σας υποστήριξη. Είναι μια ανηφόρα που πρέπει να την ανέβουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε όλα τα προσόντα για να συνεργαστούμε σωστά και να τα καταφέρουμε. Και κάτι τελευταίο είναι ότι ο πρόεδρος έκανε αυτή την, αυτό το διακανονισμό, οπότε ο πρόεδρος δείχνει σαφή δέσμευση για το θέμα της ανάπτυξης. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι παλαιότερα, όπου ο Επίτροπος της ε, Ανάπτυξης είχαν ένα, είχε ένα τμήμα μόνο πολιτικής, δεν μπορούσε να επηρεάζει, δεν είχε μεγάλο περιθώριο ελιγμών και δράσεις, οπότε νομίζω ότι τώρα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα υπό αυτές τις συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για να τη χρησιμοποιήσουμε. Το πώ θα τη χρησιμοποιήσουμε βέβαια εξαρτάται από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω να τη χρησιμοποιήσω με, το καλύτερο, με τον καλύτερο τρόπο. Μην με κρίνετε όμω από την πρώτη εβδομάδα. Είναι πολύ νωρί ακόμη να ε, πείτε αν τα πάω καλά ή άσχημα. Εγώ σα είπα ότι αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη ενώπιον τη Επιτροπή σα και όποτε επιθυμείτε μπορώ να έρθω εδώ να σα ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εντάξει, και εσείς δεν ήσασταν σοφοί όταν πρώτο ξεκινήσατε. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα είναι απολύτω διαφανή τα πράγματα και ελπίζω να καταλήξω στα επιθυμητά αποτελέσματα. Thank you. Mr. Deva has asked. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέβα ζήτησε το λόγο και νομίζω ότι είναι τελευταία ομιλητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Θέλω να σας συγχαρώ και να σας καλωσορίσω. Θα ήθελα ε, να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι μπορούμε να συμμεριστούμε απόψεις και φιλοσοφίες. Καλό θα ήταν να ξαναγυρίσουμε στα βασικά. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Ε, έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές ε, έννοιες που είναι πολύ παλιές. Συμπληρωματικότητα, συνοχή, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα, όλα αυτά μας έρχονται εύκολα. Όμως αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς η Ευρώπη έλυσε το πρόβλημα της φτώχειας, οι Ηνωμένε Πολιτείε πώς ξέφυγαν από τη φτώχεια ή πώς 300 ε, εκατομμύρια Κινέζοι ε, μείωσαν το επίπεδο της φτώχειας, βελτίωσαν τη ζωή τους αν θέλετε. Η διαδικασία δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη, αλλά τη δημιουργία πλούτου, ευημερίας. Η κυρία Τζόλι μας έδειξε πολύ αποτελεσματικά ότι περίπου 800 δις ευρώ έρχονται από τις αναμνησόμενες χώρες, ενώ εμείς Βάζουμε 8 δις στο κοινοτικό προϋπολογισμό και στο ΕΤΑ 23 εκατομμύρια κάθε τέσσερα χρόνια. 800 δις όμως μπαίνουν από εκεί εδώ κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για έλλειψη χρημάτων. Τα 800 εκατομμύρια βγαίνουν. Άρα αυτά τα 800 δις γιατί δεν τα αφήνουμε να χρησιμοποιηθούν στις χώρες αυτές Πώς μπορεί το χρήμα αυτό να μείνει στις χώρες αυτές. Πώς μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των χωρών αυτών στις χώρες αυτές. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ευημερία και πλούτος με το χρήμα αυτό σε αυτές τις χώρες. Δημιουργία πλούτου, γιατί κάποιες ε, αφρικανικές χώρες είναι από τις πλουσιότερες σε πρώτες ύλες στον κόσμο. Όπως ακούσαμε όμως, φεύγουν τα χρήματα. Δηλαδή τεράστιες ποσότητες νερού, και ε, χρημάτων βγαίνουν από εκεί και εμείς επιστρέφουμε μια δαχτυλίθρα. Πώς μπορεί λοιπόν να μείνουν εκεί οι πόροι αυτοί και να βοηθήσουν τις χώρες αυτές. Κύριε Πίπαγης. Έχω μικρή εμπειρία στην πολιτική ανάπτυξη. Έχω όμως κάποια εμπειρία στη διαδικασία ένταξης. Ήμουν λετονός και μπορούσα να παρακολουθήσω το παράδειγμα της χώρας μου, ξέρω όπως το καταλαβαίνω. Υπάρχει λοιπόν, υπήρξε μάλλον μια προενταξιακή περίοδος και κατά τη διάρκεια εκείνη η αντιμετώπιση δεν ήταν τόσο ε, τι θα κερδίσουμε, αλλά τι υποδομή φτιάχνεις. Διότι χωρίς υποδομή, χωρίς capacity building δεν μπορείς να φτιάξεις διακυβέρνηση. Χωρίς διακυβέρνηση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Νομίζω συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε να έχει χρειαζόμαστε να, υπάρχει, να υπάρχουν κονδύλια, αλλά χρειαζόμαστε και διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει διακυβέρνηση, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει διασπάθηση. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πρέπει να βάζουμε λίγα κονδύλια εκεί που δίνουν τις καλύτερες ευκαιρίες για την κυβέρνηση. Έτσι μόνο μπορούμε να πετύχουμε. Δεν νομίζω ότι απλώς είναι καλό να στέλνουμε κονδύλια στη χώρα ελπίζοντας ότι κάπως θα λυθεί το πρόβλημα. Και ε, με την εμπειρία της χώρας μου θα σας έλεγα ε, και να μην είχαμε γίνει μέλος της Ένωσης με τη δουλειά που είχαμε κάνει προενταξιακά θα, θα έχω, είχα εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. και η διαδικασία δεν θα ήταν τόσο εύκολη. Μην ξεχνάτε ότι ε, στην εποχή εκείνη υπήρχαν σοβαρότατες επικρίσεις για το τρόπο που δουλεύαμε. Μας λέγανε ότι δίνουμε λεφτά, τα λεφτά που παίρνουν από την Ένωση σε, σε εταιρείε συμβούλων επιχειρήσεων από τη Δύση μόνο και μόνο για να κυκλοφορούν τα χρήματα. Ωστόσο εμείς διαπιστώσουμε ότι αυτό ήταν εμπειρία. Επίσης, τα ΙΣΠΑ τα προγράμματα ΙΣΠΑ για τις μεγάλες υποδομές είχαν θεωρηθεί ως υπεργραφειοκρατικά. Αλλά μάθαμε με τα ΙΣΠΑ πώς να φτιάχνουμε εμείς, ε, να προετοιμάζουμε εμείς έργα υποδομής. Και αυτό λοιπόν ήταν ε, θετικό και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις. <coughs> merci à Monsieur le Commissaire d'être venu. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο που ήρθε μαζί μας για να μοιραστεί μαζί μας τις πρώτες εμπειρίες του από αυτή τη, νέα του θέση. Να τελειώσουμε τη συνεδρίαση. Μόνο μη φύγετε ακόμα. Θα έχουμε τη συνάντηση των συντονισμών στις 6 και 4. Των συντονιστών, συγγνώμη. Υπάρχει το σημείο διάφορα ακόμα στη μέση διάταξη. Υπάρχει κανείς Στα διάφορα έχετε κάτι? Όχι. Η επόμενη συνάντηση στις Βρυξέλλες 1η Μαρτίου 3 με 6.30 και στις 16 Μαρτίου 3 με 6,5 επίσης. 17 Μαρτίου 9 με 6,5. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση, θα γίνει συνάντηση των συντονιστών σε 5 λεπτά εδώ. Οι συντονιστές...